Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είσαστε παρόντες. Και χαίρομαι που είναι τόσοι εκπρόσωποι της νέας γενιάς εδώ. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Ξέρετε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα και το δείχνει και η παρουσία σας εξάλλου. Χαιρόμαστε γιατί έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για κάτι το οποίο για τη δική σας γενιά είναι το σημαντικότερο και είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσει. Η παιδεία, η κατάρτιση, η υπέρβαση της ανεργίας των νέων. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι πολλά αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά έχουμε πολύ μεγάλες στενοπούς χρηματοδότησης σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό όταν επίσης η Κομισιόν θέλει να ενισχύσει τα προγράμματά της, δεν ξέρουμε από πού θα βγουν τα λεφτά αυτά. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι σαφέστερα τα κονδύλια που θα δοθούν για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε με σοφροσύνη. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν καταλαβαίνουν ότι οι περικοπές στην εκπαίδευση φέρουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο θέλουν να επιτύχουν. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα της Ευρώπης 20%. Θέλουμε να μειώσουμε το ποσοστό σχολικής αποτυχίας. Θέλουμε να φτάσουν αυτοί οι οποίοι τελειώνουν το πανεπιστήμιο, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο μάλλον στο 40% ή περισσότερο για όλα αυτά όμως χρειαζόμαστε να έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας και η Κομισιόν αυτό θέλει να επιτύχει, αλλά βρισκόμαστε ακόμα μακριά από αυτό το στόχο. Έχουμε το πρόγραμμα της διαβίου εκπαίδευσης, το οποίο προωθεί την κινητικότητα των ε, σπουδαζόντων και των καθηγητών. Έχουμε επίσης την εκπαίδευση η οποία είναι επαγγελματική, την εκπαίδευση των ε, επαγγελματικά είδη ενεργών, τα προγράμματα Λεωνάρντο, Κομένιους και για αυτούς οι οποίοι ξέρουν το πρόγραμμα Εράσμους, γιατί είναι και το παλιότερο από αυτά τα προγράμματα, μπορώ να σας πω ότι η πελατεία του Κομένιους και του Λεωνάρντο γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν με τα προγράμματα αυτά. Το Έρασμος και όλα αυτά τα προγράμματα είναι ίσης αξίας, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως ίσης αξίας και για τους νέους που είναι εδώ παρόντες, θέλω να πω ότι και η νεότης ενδράση είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Με τα στοιχεία του Alpha Tempus, Edulink, Edulink Erasmus Tempus και με τη συνεργασία με άλλες βιομηχανικές χώρες έχουμε την συνεργασία στο πανεπιστημιακό επίπεδο που ξεπερνάει πια και τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι το πρόγραμμα νεότης σε δράση πρόκειται για δράσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες για άτυπες μορφές εκπαίδευσης και θέλω επίση να υπενθυμίσω το πόσο σημαντικό είναι το, πρόγραμμα της εθελοντικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πετύχει πολλά με τη διαβίω εκπαίδευση και τη νεότητα σε δράση. Όλες οι όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε για τα προγράμματα αυτά μας δείχνουν ότι έχουμε πετύχει πολλά για τους ανθρώπους στην Ευρώπη με τα προγράμματα αυτά και η επόμενη γενιά προγραμμάτων θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα διδάγματα αυτών των προηγουμένων προγραμμάτων και να βασιστεί σε αυτά ώστε να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες όλων αυτών που χρειάζονται υποστήριξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Έχουμε σήμερα λοιπόν μια ακρόαση με εκπροσώπους από, διάφορες, από διάφορες τομείς εκπαίδευσης. Χαίρομαι για την παρουσία του, του δόκτωρα Τόμας Σπίλκαπ, ο οποίος είναι ο ασκόντα καθήκοντα του διευθυντού της Pädagogischer Austauschdienst στη Γερμανία, της υπηρεσίες δηλαδή για παιδαγωγικές ανταλλαγές. Και έχουμε επίσης ένα εκπρόσωπο του Φόρουμ των Νέων, τον Πέτερ Ματσιασικ, από το Βέλιο Το όρμα βέβαια δείχνει ότι έρχεται κάπως μακρύτερα από το Βέλιο Έχουμε μετά τον κύριο Βούτιχ, ο οποίος είναι ο διευθυντής της DAD, της ε, Γερμανικής Ακαδημίας Ανταλλαγών, Ακαδημαϊκών Αλλαγών μάλλον, και τον κύριο Ζάλμπερκ, Πάζη Ζάλμπερκ, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Κέντρου για Διεθνή Κινητικότητα από τη Φιλανδία. Η ακρόαση τώρα είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε θα έχουμε καταρχήν ένα γύρο παρουσιάσεων από τους ομιλητές μας, περίπου 15 λεπτά ο καθένας. Θα ακολουθήσει ένα τμήμα όπου για μία ώρα θα μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις και θα έχει 5 με 10 λεπτά ο καθένας από τους ομιλητές χρόνο για να απαντήσει στα ερωτήματα. Στο τέλος θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Κορσέλ, να λάβει το λόγο, να μας αναφέρει ποια είναι η άποψή του για αυτά τα οποία έχουν ακουστεί εδώ. Να σας πω επίσης και για ορισμένα τεχνικά θέματα. Η συνάντηση αυτή βρίσκεται, μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Ό,τι και να κάνετε λοιπόν, άμα καθαρίζετε τη μύτη σας ή τα αυτιά σας, αυτό θα φανεί στο διαδίκτυο. Για να είσαστε στην εικόνα όταν ομιλείτε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο το οποίο βρίσκεται ε, δεξιά σας. Έρχομαι τώρα λοιπόν στην ακρόαση και δίνω καταρχήν το λόγο στον κύριο Σπίλκαμπ ο οποίος θα αναφερθεί κυρίως στο θέμα των σχολείων και τη σημασία του Κομένιους και των νέων προγραμμάτων για τα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζετε εξάλλου ότι στις ε, χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη και εκεί μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σπίλκαμπ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να σας γυρίσω την πλάτη σε ορισμένου από εσά. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα κάνει λιγότερο ενδιαφέρουσα την παρουσίασή μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε στην Επιτροπή Πολιτισμού και ε, Εκπαίδευσης. Είναι μια μεγάλη τιμή να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε την απόψή μας εξ ονόματος των διδασκόντων στα σχολεία. Αργαζόμαστε εδώ και 60 χρόνια με το πρόγραμμά μας στη Γερμανία για ανταλλαγές με 90 ε, χώρες του κόσμου και αυτό δίνει τη δυνατότητα στη μαθητιώσα νεολαία να έχει τις δυνατότητες αυτών των ε, ανταλλαγών. Θα μιλήσω τώρα και για τα θετικά και για, τα, για, τους κινδύνους των προγραμμάτων αυτών με, το, με την ακροστιχιδα Κομένιους. Έχουμε καταρχήν τις ανησυχίες για το Εράσμους για όλους, τις υποχρεώσεις του προγράμματος αυτού για το σχολικό τομέα, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή αυτών που κάνουν αίτηση, να έχουμε καλύτερη δίκηση, να συμπεριλάβουμε όλα τα σχολεία, να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αντίκτυπο, να συνδυάσουμε διαφορετικούς τομείς ε, παιδείας και να ενισχύσουμε το σχολικό τομέα. Αυτό είναι και το συμπέρασμα στο οποίο θέλω να καταλήξω. Οι ανησυχίε μα σε σχέση με το πρόγραμμα διάδοχο, το Έρασμο για όλου. Από το ε, ε, από δεκαετία 1960 το Έρασμος είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το Κομένους βέβαια είναι νεότερο στην ηλικία πρόγραμμα και δεν είχε τη χρηματοδότηση του Εράσμου. Το Κομένους έχει σαν στόχο την καινοτομία στο σχολικό τομέα. Όταν υπάρχει το όνομα Κομένιους δίπλα στο όνομα ενός σχολείου, ξέρουν όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το πρόγραμμα αυτό, τους δίνει μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Οι σχολές και οι μαθητές συνδέουν σήμερα την Ευρώπη μέσω με το Κομένιους. Συνδέονται μέσω του Κομένιους. Είναι για ορισμένους όχι ιδιαίτερα εύκολα καταλάβει κανείς τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα αυτό και γι' αυτό πρέπει να σταθώ στο θέμα αυτό. Είναι τρεις οριζόντιες δράσεις που θέλουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή στο νέο πρόγραμμα Έρασμος για όλους και αυτό ίσως είναι πολύ απλοποιημένο για μια πολύ πολύμορφη και πολύπλοκη πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Με το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα έχουμε το πρόβλημα ότι αναμειγνύουμε τελείως διαφορετικές ομάδες στόχους. στόχου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ των ε, σχολείων και των, ε, των μικρών σχολείων ή των μεγάλων και των πανεπιστημίων, δηλαδή πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση η οποία είναι ειδική κατά τομέα. Από την πλευρά των σχολείων αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ασαφές και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή στην οποία παίρνουν οι διάφορες δράσεις. οι υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατά την άποψή μου είναι να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ομάδων στόχου. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη ή τη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο στόχος είναι να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των χρηστών των προγραμμάτων. Γιατί όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτά τα προγράμματα εργάζονται και πέραν του χρόνου εργασίας τους, του κανονικού χρόνου εργασίας τους αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια πίεση πάνω στα σχολεία, είναι υποχρεωμένα να μειώσουν τις δαπάνες τους και όχι να τις ενισχύσουν. Τα σχολεία θα πρέπει να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συγκεκριμένες ανάγκες για δράσεις. Θέλουν να έχουν καλύτερη αμοιβαία γνώση, να υπάρξει μεταλαμπάδευση διδακτικών μεθόδων και καλύτερη συνεργασία με άλλα σχολεία. Δηλαδή, τα σχολεία θέλουν μια απλή προσέγγιση. Μια μη γραφειοκρατική αντιμετώπιση και μη γραφειοκρατική προσέγγιση στα προγράμματα αυτά. Ο στόχος τους είναι καταρχήν το να μπορέσουν να διαπαιδαγωγήσουν τις επόμενες γενιές και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να παίξουν ένα πρόσθετο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να είναι πιο εύκολη η ζωή αυτών οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια αίτηση για τα προγράμματα αυτά. Με συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουμε όλες τις δράσεις οι οποίες μέχρι τώρα ήταν μέσα στο κομμένιος, αλλά να τις απλοποιήσουμε. Θα πρέπει να μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνονται αιτήσει με μια λογική μενού, όπου υπάρχουν ελκυστικές προτάσεις για τους διδάσκοντες, για τους διδασκόμενους, και να μπορεί κανείς να επιλέξει από αυτούς ακόμα και να προβλέπεται η μακροχρόνια κινητικότητα για τους ε, μαθητές. Τώρα για τους ε, καθηγητές ίσως δεν είναι απαραίτητη μια τέτοια μακροχρόνια ε, κινητικότητα. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε σταματήσει αυτό το πρόγραμμα για τους διδάσκοντες γιατί ούτως ή άλλως ήταν πολύ μικρή ζήτηση γι' αυτό. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια δράση που αφορά τους επικεφαλείς των σχολείων, παραδείγματος χάρη ανταλλαγές επισκέψεων κτλ. Δεν έχει νόημα να συναντούν μονάχα οι επικεφαλής των σχολείων μόνο επικεφαλής άλλων σχολείων. Αυτό δεν τους εμποδίζει να αναπτύξουν μια ευρύτερη προοπτική σε σχέση με τα σχολικά προβλήματα. Πρέπει παράλληλα να μειωθεί η γραφειοκρατία στα νέα προγράμματα, να μείνει σε ένα ελάχιστο επίπεδο Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιβαρύνουμε τους αποδέκτες των προγραμμάτων με πρόσθετη γραφειοκρατία. Επομένως, ε, εν γέννη τα σχολεία της Ευρώπης δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μεγάλα ευρωπαϊκά σχέδια και να αναλάβουν την ε, δημοσιονομική ε, ευθύνη, παραδείγματος χάρη, για να μεταφέρουν κονδύλια σε άλλα σχολεία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο τους έρχεται εύκολο. Πώς μπορούμε τώρα να έχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση των νέων προγραμμάτων, ένα θετικό στοιχείο για την τωρινή γενιά προγραμμάτων είναι η δυνατότητα να γίνονται εταιρικέ σχέσεις περιστασιακά για σύντομα χρονικά διάστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί και στο μέλλον. Έχουμε αρνητικά, προ... στοιχεία όταν στο Κομένιους Ρέγγιο υπήρξαν κάποιες ε, διατάξεις οι οποίες ήταν πολύ περιοριστικές, οι ίδιες διατάξεις διαχείρισης που είχαν να κάνουν με τεράστια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτρέπει βέβαια την ε, αξιοποίηση προγραμμάτων στα οποία μπλεκόσασταν μονάχα μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση του προγράμματος, των προγραμμάτων αυτών, πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη διοικητική ικανότητα στους εθνικούς φορείς. Επομένως, ένα μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού για τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να έχει και εθνικό χαρακτήρα, και να δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθούν οι απαραίτητες διοικητικέ δομές σε εθνικό επίπεδο. Μια βελτίωση στη διαχείριση θα ήταν να υπάρξει και μεγαλύτερος ρόλος των εθνικών ε, φορέων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ιδιαίτερη ορατότητα αυτών των φορέων το να παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο θα μπορούσε να ενισχύσει ιδιαίτερα αν υπάρξει και η υπευθυνοποίηση των εθνικών φορέων. Επίσης, πολύ σημαντικό για τα θέματα αυτά είναι να υπάρξει μια συνεχής παρακολούθηση από τους εθνικούς φορείς σε σχέση με το περιεχόμενο και εκεί πρέπει να υπάρξει έμφαση και όχι μονάχα σε μια διοικητική δημοσιονομική διαχείριση. Θα πρέπει λοιπόν στο επόμενο πρόγραμμα να τεθεί η έμφαση στο περιεχόμενο και την ποιότητα και θα πρέπει να αποφύγουμε ε, επαχθείς διαχειριστικές δομές οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με, το, με τους στόχους του πραγματικούς του προγράμματος αυτού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να θεωρήσουν ότι εμπλέκονται από αυτό το πρόγραμμα, ότι τα προγράμματα αυτά είναι προς όφελος των ομάδων στόχου και όχι μόνο της διοίκησης, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τα παλιά σχολεία, <clears throat> αυτά που έχουν πείρα στα προγράμματα αυτά, και τους νεοφερμένους και τα μικρά σχολεία και τα μεγάλα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις και τα σεμινάρια επαφής. Μπορεί να είναι πολύπλοκα σε επίπεδο διαχείρισης, αλλά με τον τρόπο αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα σχολεία να γνωρίσουν αυτά τα προγράμματα. Επίσης, κατά τη δική μου άποψη, χρειαζόμαστε και μικρής κλίμακος σχέδια, ακόμα και απλά διμερή σχέδια. Όταν δεν υπάρχουν αρκετοί ε, εταίροι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Και επίσης μπορεί ένα σχολείο να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα μονάχα και για ένα σχολικό έτος και όχι παραπάνω, εφόσον το επιθυμούν. Από τη δική μου εμπειρία Νομίζω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να καλύπτονται να καλύπτονται τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των ομάδων ε, στόχου. Επίσης πρέπει να αυξήσουμε τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα στα νέα αυτά προγράμματα, κάτι το οποίο εδώ παίζει σημαντικό ρόλο είναι η καλύτερη διασύνδεση των προγραμμάτων αυτών με την πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δεν μπορεί κάθε πρόγραμμα σε σχολικό επίπεδο να επιτύχει τη μείωση του ποσοστού αυτών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Θα πρέπει να είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχουν προγράμματα τα οποία δεν συνδέονται ένα προς ένα με τα σχέδια, με τους στόχους παραδείγματος της Ευρώπης 2020. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια πιο θεσμική αντιμετώπιση όταν πρόκειται για τη συνεργασία προς την κατεύθυνση ενός συγκεκριμένου στόχου και να μην θεωρείται ότι μονάχα εξυπηρετούμε ένα περιστασιακό στόχο. Πολλά αυτά τα οποία ε, γίνονται με τα προγράμματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή μιας σχολικής κοινότητας, αλλά ιδίως και για τη ζωή των <clears throat> διδασκομένων τε και διδασκόντων. Δεν είναι πάντα καταμετρήσιμη βέβαια αυτή η επίδραση και ο αντίκτυπος. Φαίνεται μονάχα μετά από πολλά χρόνια και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει, να πριτανεύσει η αρχή της εμπιστοσύνης για τα προγράμματα αυτά, γιατί πάρα πολλά θετικά γίνονται με αυτά τα προγράμματα, ακόμα και δεν είναι άμεσα καταμετρήσιμα. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, κυρίως με την ενισχυμένη παρουσία των διδασκόντων, και θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα και όχι να την υποβάλουμε σε επαχθείς διαδικασίες υποβολής προτάσεων. Επίσης μια άλλη σημαντική ιδέα είναι η ηλεκτρονική αδελφοποίηση των σχολείων μέσα στο σχολείο αυτό. Να έχουμε δηλαδή σχέδια μέσα στα οποία μπορεί να υπάρξει η αναζήτηση εταίρων μέσα από τα οποία επίσης μπορεί να υπάρξει και μία πρόοδος σε σχέση με τις σχολικές πολιτικές και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με τη βοήθεια του διαδικτύου. Θέλω να τονίσω τώρα τη σημασία του να διασυνδέσουμε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς. Η βασική ιδέα του σχεδίου είναι βέβαια σωστή ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ τομέων και να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ τους. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο πυρήνας του νέου προγράμματος. Πιστεύω ότι ο κάθε τομέας έχει τις δικές του ανάγκες. Ο καθένας είτε είναι μαθητής είτε είναι ε, φοιτητή στο πανεπιστήμιο είτε είναι πανεπιστημιακός είτε διδάσκω σε σχολείο έχει διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετικό στόχο. Επομένως μια προσέγγιση κατά θα είναι πιο αποτελεσματική και θα ενισχύσει τον αντίκτυπο αυτού του προγράμματος. Ένα καλό παράδειγμα είναι τα τωρινά προγράμματα Comenius Regio, όπου έχουμε μια προσέγγιση η οποία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αποτελέσει και υπόδειγμα. Εξασφαλίζει μια καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναπτύξουμε περισσότερο. Έχουμε τώρα στα συμπεράσματα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των σχολείων εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Ο σχολικός τομέας δεν είναι μονάχα η βάση της οποιασδήποτε γνώσης, αλλά έχει την μεγαλύτερη ομάδα στόχου αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρώπη. Η στρατηγική για την νεότητα σε δράση δεν έχει αντιμετωπίσει αρκετά την ε, προβληματική της ε, μαθητιώσας νεολαίας και φοβάμαι ότι και το νέο πρόγραμμα μπορεί να μην το πράξει. Φυσικά πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αύξηση του προϋπολογισμού για το σχολικό τομέα και αυτό θα βοηθήσει σε μελλοντικό επίπεδο την Ευρώπη. Τέλος, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε την διαδικασία αυτή που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης. Θέλουμε να ξέρουμε ότι ο κάθε μαθητής θα ξέρει τι είναι η Ευρώπη, τι οφείλει στην Ευρώπη και θα μπορέσει με τον τρόπο αυτό να γίνει ένας ενεργός και υπεύθυνος Ευρωπαίος πολίτης. Και τέλος θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης ξεκινάει την ενεργή του ζωή σαν μαθητής στο σχολείο. Και σας υπενθυμίσω τώρα κλείνοντας τη συζήτηση που είχα στη Βαρσοβία με ένα Πολωνό δάσκαλο σε μια συνδιάσκεψη στη Βαζοβία. Αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτό που είπε. Μου είπε ότι ότι τα πρώτα πράγματα που είδε γραμμένα είχαν γραφτεί από τη γιαγιά του και έλεγε, έλεγαν θάνατος. Ο θάνατος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου του 1939. Στο σχολείο λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να γίνονται σαφή στους μαθητές, οπότε αυτό το παράδειγμα ήταν ένα παράδειγμα με το οποίο μπορούσε να δείξει στους μαθητές του ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι κάτι το δεδομένο, δεν είναι κάτι το προφανές. Κάθε νέα γενιά πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οδήγησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόγραμμα διάδοχος, το Έρασμος για όλους, θα πρέπει να λάβει υπόψη σημαντικότερα τα θέματα του σχολείου και θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα Κομμένιους έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμή μια μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Συνεχίζουμε τώρα με το πρόγραμμα Νεότης σε δράση και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάτια Σικ ο οποίος έχει και αυτός να κάνει μία παρουσίαση ισχυρού σημείου. Δεν έχετε PowerPoint. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να λάβετε το λόγο και να συνεχίσετε. Σας δίνω το λόγο παρ' όλα αυτά. Είσαστε ο νεότερος εμπειρογνώμων εξάλλου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, και αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι, βρίσκομαι εδώ σήμερα ως ε, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, ενός φόρουμ που εκπροσωπεί 98 διεθνείς ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, από προσκόπους μέχρι οργανώσεις φοιτητών, από την Ισλανδία μέχρι το Αζερμπαϊτζάν, από την Πορτογαλία μέχρι τη Φιλανδία. Εκατομμύρια νέων λοιπόν... Λίγο, πιο αργά λέει και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μοιραστούμε μαζί σας ε, την εμπειρογνωμοσύνη μας ε, σε ό,τι αφορά το ε, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Νεολαία. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε σήμερα ένα τέτοιο συνεχές πρόγραμμα αντί για ένα Εράσμου για όλους. Γιατί αυτό το μελλοντικό πρόγραμμα θα ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, της των νέων μορφών εργασίας, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι και θα, μας, τους βοηθήσει να μετατραπούν ε, και να διαμορφωθούν σε ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες. Η πρόταση Erasmus for All ε, οδεύει προς σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στη μάθηση και την έμφαση στην ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και τον εθελοντισμό. Ωστόσο, δεν ε, έχει ικανοποιητικές λύσεις σε ό,τι αφορά τις ε, ανάγκες όλων των ε, νέων σε επίπεδο αναγνώριση της εργασίας των νέων, σε οργανώσεις νεολαίων για την στήριξη της αυτονομίας των νέων. Το ανανεωμένο αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα εστιαζόμενο στις ε, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της μη επίσημης, ανεπίσημης ε, εκπαίδευσης, συμμετοχής και του εθελοντισμού. Στην παρουσίασή μου εγώ θα σας παρουσιάσω κάποια επιχειρήματα, επιχειρήματα που εξηγούν γιατί κατά τη γνώμη μας η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής δεν είναι Απολύτω ικανοποιητική και γιατί μετά από τι διαβουλεύσεις ε, που έχουν γίνει εμεί ε, επιμένουμε στο αίτημά μα για ένα νέο και ανεξάρτητο ε, πρόγραμμα για την νεολαία σε δράση. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Νεότητα θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ε, να, να καταστήσει την πολιτική για την νεολαία της πολιτική και οικονομική, δημοσιονομική προτεραιότητα. Σήμερα μέσα στην κρίση οι επενδύσεις, το να επενδύσουμε στην νεολαία θα αυξήσει την κοινωνική συνοχή και, και γι' αυτό εμείς χαιρετίζουμε την έμφαση που δίνεται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, στον, στην κινητικότητα των νέων, την ε, άτυπη επίσημη και ανεπίσημη ε, ε, εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και το καθεξής και στηρίζουμε την αύξηση της χρηματοδότησης αυτού τους τομείς. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι το Youth in Action έχει νόημα και από δημοσιονομικής πλευράς. Σε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα, σε έκθεσή του υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα ε, νεολαία στην ε, ε, νεολαία σε δράση έχει χαμηλό κόστο ως αναδικαιούχο και γι' αυτό είναι και ιδιαίτερα αποδοτικό. Και αυτό συνδέεται και με την έκκληση του κυρίου Μπαρός ότι κάθε ευρώ που θα ξοδεύεται μέσα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει αξία και νόημα το European Youth Forum έχει ζητήσει αυτό το ανεξάρτητο πρόγραμμα να συνεχιστεί και μετά το 2013. Όμως αυτό δεν φαίνεται τώρα στην πρόταση της Επιτροπής για το Εράσμους για όλους. Εμείς επικαλούμεθα τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για το ε, πρόγραμμα αυτό, όπου πάνω από 7.000 ε, άτομα, φορείς ε, και δημόσιοι φορείς συμμετείχαν. 40% αυτών ήταν υπέρ της συνέχισης της εφαρμογής του προγράμματος ξεχωριστά και και 43% είπαν ότι το, θα πρέπει να, το, τα προγράμματα να υλοποιούνται ξεχωριστά, αλλά με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν και με τη θέση πολλών κρατών μελών που έχουν ζητήσει τη διαφοροποίηση, ε, του προγράμματος. Το ίδιο αναφέρθηκε και σε μια ε, συνδιάσκεψη για την νεότητα της ε, Δανικής Προεδρίας και στις κοινέ του συστάσεις ε, αναφέρεται ότι οι νέοι χρειάζονται έναν ανεξάρτητο μηχανισμό που θα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεότητα που ε, θα έχει δική της γραμμή προπολογισμού. Αυτό θα διασφαλίσει ότι και οι οργανωμένοι και οι μη οργανωμένοι νέοι και ε, οργανώσεις νέων θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα αυτό με έναν εύκολο τρόπο. Βεβαίως η μεγάλη πλειονότητα αυτών των δικαιούχων που αξιοποιούν αυτά τα κονδύλια αλλά και οι περισσότεροι αξιωματούχοι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι είναι υπέρ ενός ανεξάρτητου και ξεχωριστού προγράμματος. Αυτή η δημοκρατική φωνή προς το παρόν αγνοείται από το ε, την τρέχουσα πρόταση και απορρίπτεται από την Επιτροπή. Γι' αυτό και εμείς ε, ως εκπρόσωποι ε, των Ευρωπαίων πολιτών απευθυνόμαστε σε εσά. Τι θέλει λοιπόν αυτό το φόρουμ. Εμείς ζητήσαμε ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να να αποτελέσει ένα μέσο με το οποίο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της βάσει της ε, συνθήκης της Λισαβόνα, ιδιαίτερα του άρθρου 165, για την ε, συμμετοχή ε, των νέων στην Ευρώπη. Τέτοια άρθρα στο παρελθόν οδήγησαν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν τη Ευρωπαϊκή για την Νεολαία θα πρέπει να αποτελέσει ένα εργαλείο για την υλοποίηση του συμπληρωματικού πολιτικού θεματολογίου, το πλαίσιο για την ε, στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ε, νεότητας. Θέλουμε ένα πρόγραμμα που να εστιάζει στην ε, ανεπίσημη εκπαίδευση των νέων, στην, στην εργασία και έτσι να στηρίζουμε την αυτονομία των νέων μέσω ενός ευρέως φάσματος οργανώσεων νέων που εκπροσωπεί πάρα πολλού νέου στην Ευρώπη. Γιατί το θέλουμε αυτό. Εξαρτάται από το τι θέλουμε για ένα, από ένα μελλοντικό πρόγραμμα. Κατά τη γνώμη μα, θα πρέπει να αντιμετωπίζει και να πληρεί τι ανάγκε όλων των νέων σε όλη την Ευρώπη. Η ανταπόκριση που σημειώθηκε στι δημόσιε από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι οι μεγαλύτερε προκλήσει είναι οι κοινωνικέ αλλαγέ, ε, η ανεργία στους νέους και οι αλλαγές της ανάγκης της αγοράς, ε, ε, διακρίσεις, ρατσισμός και εξονοφοβικά φαινόμενα ε, στους νέους ε, και ο αποκλισμός των λιγότερο προνομιούχων νέων. Αν δούμε τι προκύπτει και από, τον, ε, από την αξιολόγηση αντικτύπου, βλέπουμε ότι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι νέοι και μάλλον το, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το να δώσουμε στους νέους τις απαραίτητες δεξιότητες ούτως ώστε για να τους προετοιμάσουμε για την αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς και δραματικά ε, και πλέον μεταφερόμαστε σε μια κοινωνία που βασίζεται στην γνώση. Σε αυτό λοιπόν ε, το δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό ε, πλαίσιο οι νέοι πλέον πρέπει να πληρούν πολλά περισσότερα κριτήρια με πολλές περισσότερες δεξιότητες. Και εφόσον ζουν σε ένα τέτοιο διαφοροποιημένο αλλά και γυράσκον πλαίσιο, μια τέτοια κοινωνία που πλέον μεγαλώνει, ε, απαιτείται και μια διαμόρφωση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, ενός πνεύματος αλληλεγγύης, ε, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Το πρόγραμμα Erasmus for All δυστυχώς δεν πληρεί αυτά τα κριτήρια. Οι νέοι στην Ευρώπη είναι μια εξαιρετικά ε, πολύμορφη ομάδα. Έχουν όμως μια κοινή ανάγκη, την ανάγκη να γίνουν αυτόνομοι και ανεξάρτητοι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι θα έχουν την απαραίτητη στήριξη, πόρου και δυνατότητες, ευκαιρίε, για να ζουν ανεξάρτητοι, να κάνουν μόνο του τη ζωή τους, ε, να χαίρουν πλήρου πλήρους ε, και πολιτικής συμμετοχής σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής και να είναι σε θέση να ε, λαμβάνουν τι αποφάσει του ανεξάρτητα τα, συστήματα, επίσημα συστήματα εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν αυτά τα, ζητήματα, αλλά δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μόνοι του. Το, η ενδιάμεση εξελόγηση του Youth in Action έχει δείξει ότι εστιάζει την προσοχή του στην, στα επίσημα ε, συστήματα, αλλά θα πρέπει να δρά συμπληρωματικά ως προς τα υπόλοιπα. Κάτι άλλο το οποίο φάνηκε από τι διαβουλεύσει είναι η προστεθέμενη αξία του Youth Forum, γιατί οδηγεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ε, όπω περισσότερο από κάθε άλλο ε, μέσο. Και συμβάλλει στην ε, ανάπτυξη των τέτοιων οργανώσεων νέων περισσότερο από κάθε άλλο φορέα. Ωστόσο, ο χαρακτήρας αυτών των στοιχείων τα οποία μετράμε, που είναι δύσκολα να αποστοκοποιηθούν, καθιστά δύσκολη και την τον των αποτελεσμάτων της, όπως για παράδειγμα στην ε, επίσημη εκπαίδευση. Με την ε, διάδραση στο τοπικό περιβάλλον, ε, οι νέοι αποκτούν πολλές νέες δεξιότητες. Αλλά τι είναι ακριβώς αυτές τις δεξιότητες, η ομαδική εργασία, η αυτοπεποίθηση, η πειθαρχία, η ευθύνη, η υπευθυνότητα, ε, ο ηγετικός χαρακτήρας, ο προγραμματισμός, ε, η οργάνωση, ο συντονισμός και ε, δεξιότητες επίλυσης πρακτικών προβλημάτων. Η ανεπίσημη λοιπόν εκπαίδευση μπορεί να δώσει δυνατότητα στους νέους να συστήσουν τα δικά τους προγράμματα όπου έχουν κεντρικό ρόλο Να αποκτήσουν λοιπόν όλε αυτέ τι δεξιότητε τη αυτοπεποίθηση, τη πειθαρχία κτλ. Και έτσι να αποκτήσουν δεξιότητε στην πράξη. Και αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά ω προ τι δεξιότητε που λαμβάνουν από τα επίσημα συστήματα. Ε, και, όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο και της διαβίου μάθησης, όπου βλέπουμε ότι όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά. Εμείς χαιρετίζουμε την ε, διαφάνεια και την προβολή της διαβίου ε, ε, εκπαίδευσης μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά η απουσία της ανεπίσημης εκπαίδευση δημιουργεί πρόβλημα. Έχουμε ε, την διαβίου εκπαίδευση, αλλά δεν δίνουμε έμφαση στις οργανώσεις νέων ως ε, παρόχων ανεπίσημης εκπαίδευσης. Αυτές οι οργανώσεις είναι οργανωμένες και παρέχουν διδακτικό έργο παράλληλα με το επίσημο σύστημα εκπαίδευσης κάθε χώρας και δεν οδηγούν σε μια πιστοποίηση. Λειτουργούν επί εθελοντικής βάσης και έτσι το άτομο συμμετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία. Στην επίσημη εκπαίδευση η πάροχη είναι ξεκάθαρη. Αλλά και εδώ είναι ξεκαθαρά τα πράγματα. Οι ίδιοι οι νέοι συνέρχονται και συνεργάζονται με οργανώσεις νέων που ε, συνεργάζονται μαζί τους, ε, οι ίδιοι τις συστήνουν και παρέχουν τέτοιε δυνατότητε επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση. Οι οργανώσει νέων είναι οι πιο αποτελεσματική και αποδοτικοί φορεί ε, για την συνδρομή προ τέτοιου νέου, ιδιαίτερα του λιγότερο προνομιούχου. παρέχουμε λοιπόν ε, μακροπρόθεσμες ε, δυνατότητες εκπαίδευσης ε, και διασφάλιση βιώσιμων αποτελεσμάτων. Αυτό επιτρέπει με τη σειρά του την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Και η ενδιάμεση αξιολόγησή μας υποστηρίζει όλα αυτά τα στοιχεία. Το Youth in Action έχει μεγάλο αντίκτυπο στους συμμετέχοντες, που, που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτές τις δραστηριότητε ε, και ενισχύουν και την κινητικότητα. Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Το μελλοντικό πρόγραμμα λοιπόν θα πρέπει να βασίζεται και να οικοδομεί πάνω σε αυτή τη βάση και και όλα αυτά για να παρέχουμε ακόμα περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση, περισσότερες δυνατότητε και ευκαιρίε επίσημη και ανεπίσημης εκπαίδευση ε, να τους επιτρέψουμε να δοκιμάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, να τους δώσουμε το χώρο να συμμετάσχουν ε, όπου θέλουν να συμμετάσχουν εθελοντικά και να τονίσουμε και τα, τα ωφέλη της κινητικότητας στη μάθηση. Η αξιολόγηση επίσης επισημαίνει την έλλειψη δυνατοτήτων για τους νέους εργαζομένους να αποκομίσουν εμπειρίες από διαφορετικές προσεγγίσεις ε, σε ό,τι φορά για παράδειγμα το peer-to-peer -peer, to peer απο ε, από συναδέλφους τους, για παράδειγμα αξιολόγηση. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν θα πρέπει ε, να βελτιώνει τη δυναμική και την ποιότητα ε, τέτοιων οργανώσεων. Προκειμένου να κάνει κάτι τέτοιο το πρόγραμμα, θα πρέπει να δημιουργήσει περισσότερε δυνατότητε για του νέου εργαζομένου και του επιπληρωμή και του εθελοντέ, για να αναπτύξουν τι ε, μεμονωμένε του ε, και ατομικέ του δεξιότητε, αλλά να βοηθήσει και να στηρίξει και τι ε, οργανώσει νέων. Το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά το. Σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο, μόνο 43% είπαν ότι ξέρουν τι σημαίνει ακριβώ να είναι κάποιο Ευρωπαίο πολίτη και μόνο 32% είπαν ότι γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά του στου Ευρωπαίων πολιτών. Οι Ευρωπαί... Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Νέων και NGOs συμμετέχουν ε, ενεργά σε αυτή τη διαδικασία ευαισθητοποίηση του κοινού με την υλοποίηση, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ε, και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω ε, μεγαλύτερων δημοσίων διαλόγων. Αυτές οι οργανώσεις λοιπόν στηρίζουν την συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και νέων στην ευρωπαϊκή ζωή. Πρέπει λοιπόν και εμείς να τη στηρίξουμε. Το πρόγραμμα Erasmus for All δεν παρέχει ε, υποτροφίες για ή κάποια άλλα κονδύλια για, για τις οργανώσεις νέων και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η Επιτροπή όμως είναι διατεθειμένη να τους βοηθήσει μέσω project funding, χρηματοδότηση προγραμμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί αυτές οι οργανώσεις δεν κάνουν μόνο προγράμματα και projects, ε, συμβάλλουν στις πολιτικές Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και τα συνδέουν όλα αυτά με την πραγματικότητα συμμετέχουν στον διαθροτικό διάλογο που λαμβάνει η χώρα στην κοινωνία των πολιτών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πρέπει να κάνουν και προγράμματα παράλληλα, τότε θα είναι πολύ λιγότερο οικονομικά αποδοτική η δράση τους. Αυτό έχει, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και στους υπαλλήλους τους και στην ποιότητα των αποτελεσμάτων τους. Εμεί καλούμε τα ευρωπαϊκά όργανα στον κανονισμό να επισημάνουν συγκεκριμένα τη στήριξη προ αυτέ τι οργανώσει μέσω συγκεκριμένη δράση. Κάτι το οποίο ισχύει ήδη σήμερα. Πρόσφατα υπόθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παράσχει συνεχιζόμενη και βιώσιμη χρηματοδότηση για αυτές τις οργανώσεις. Α είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Θέλουμε να διατηρήσουμε το πρόγραμμα Youth in Action ω χωριστό πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να το διατηρήσουμε ω έχει. Θα πρέπει να, ε, ε, να ικανοποιήσουμε τις, ε, και αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που υπάρχουν, αλλά να άρουμε και τα εμπόδια. Πολλέ φορέ υπάρχουν διαδικασίε διπλασιασμού και επικαλύψεων μαζί με το διοικητικό άχθο τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυστηρέ και διαφανεί διαδικασίε, όμω εμεί πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία ε, και έτσι και να, να δαπανάτε το δημόσιο χρήμα, αλλά και να συμμετέχουν οι αρμόδιοι ε, φορεί. Αλλιώ τα προγράμματα αυτά θα είναι μόνο για του εμπειρογνώμονε και όχι για του πολίτε. Δεν έχω πολύ χρόνο. Κάτι τελευταίο μόνο. Οι δράσει του μελλοντικού προγράμματο θα πρέπει να ελοποιούνται από οργανώσει νέων που μπορούν να ικανοποιήσουν τι ανάγκε ε, των ε, νέων μέσω των σωστών διαδικασιών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη ε, βιώσιμων αποτελεσμάτων. Θα πρέπει και ο χρόνος ε, ε, εθελοντικής εργασίας να θεωρείται επιλέξιμο κόστος, επιλέξιμη δαπάνη. Το τρέχον πρόγραμμα Youth in Actions στήριζε τις οργανώσεις νέων γιατί ο αντίκτυπο του Youth in Action στους νέους είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να είναι και περήφανοι για αυτό το πρόγραμμα, αλλά και φιλόδοξοι. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των νέων στο δημοκρατικό βίο, να αναγνωρίζει ότι οι οργανώσει νέων είναι απαραίτητη δίωδος ε, ε, για την συμμετοχή των ε, νέων στο δημόσιο βίο και για την διαμόρφωση μιας ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνία χωρί αποκλεισμού. Και αυτό είναι η Ευρώπη που μα αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πίτερ. Ο καθηγητής Βούτιχ τώρα για τον έρασμο. Όχι για τον... Ναι, για, τον έρασμο για όλους. Δόκτωρ Βούτιχ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου της παρέμβασής μου. Καταρχήν, μια επισκόπηση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε για το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια, γιατί αυτό με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το θέμα των πανεπιστημίων, ότι έχουμε επιτύχει, που υπάρχουν ακόμα ανάγκες βελτίωσης και στη συνέχεια θα έρθω στα σχόλιά μου για την πρόταση της Κομισιόν και φυσικά και θα διεξέλθω και το θέμα του σε ποιο βαθμό αυτή η πρόταση καλύπτει τις ανάγκες της τωρινής κατάστασης και αν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συγκυρίες στις οποίες βρισκόμαστε και θα καταλήξω στο τέλος σε πέντε συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ έχετε μια ε, ταχεία επισκόπηση για τα διάφορα ε, πολιτικά μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση που εκτείνονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο και βλέπετε ποια είναι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με αυτά και ποιοι είναι οι πολιτικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Αν επανέλθουμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της Ευρώπης, την ε, ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κυρίως καλύπτεται από το πρόγραμμα Εράσμου, το οποίο γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια. Όπως βλέπετε, έχει καταγάγει σημαντικές επιτυχίες. Περίπου 3.000 πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν στην Ευρώπη, 2,5 εκατομμύρια φοιτητέ οι οποίοι έχουν μετακινηθεί με το πρόγραμμα Εράσμους, 300.000 διδάσκοντες, και διοικητική πάλι των πανεπιστημίων, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, για να εξασφαλίσουμε πιο βιώσιμα και αηφόρα στοιχεία. Δεν αφορά μονάχα τα άτομα, αλλά έχει και θετικό αποτέλεσμα για τα πανεπιστήμια, για τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και για το σύνολο της Ευρώπης. Και τέλος, αλλά όχι και το ο είναι ένα παγκόσμιο υπόδειγμα για περιφερειακή κινητικότητα και την ακαδημαϊκή συνεργασία ένα υπόδειγμα για όλο τον κόσμο. Πού υπάρχουν τώρα δυνατότητες βελτίωσης, πού υπάρχουν σημεία αδυναμίας. Καταρχήν, η γεωγραφική κάλυψη. Θα επανέλθω σε αυτό. Δεύτερον, θέλουμε να υπάρξει κάποιος εξυγχρονισμός των μέτρων αυτού του προγράμματος, το οποίο έχει μείνει ουσιαστικά το ίδιο εδώ και 25 χρόνια. Θα θέλαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό με στρατηγική ενατένιση για να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα, ένα μέσο παγκοσμιοποίησης των πανεπιστημίων. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, κινητικότητα των φοιτητών, να έχουν μεγαλύτερες υποτροφίες παραδείγματος χάρη και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και μία ε, βελτίωση της δίκησής του. Εδώ βλέπετε τη γεωγραφική εμβέλεια του προγράμματος. Βλέπετε ότι υπάρχει μία έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ του ευρωπαϊκού χώρου που καλύπτει 47 χώρες και του προγράμματος Εράσμους που καλύπτει μόνο 33 χώρες από τις 47. Αν θέλουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη υποστήριξη για τη διαδικασία της Μπολόνια στον ευρωπαϊκό χώρο, θα πρέπει να αυξηθεί η εμβέλεια αυτού του προγράμματος σε γεωγραφικό επίπεδο και να καλύψει ακόμα και πέρα των 47 χωρών. Για τις ε, υποτροφίες που δίνονται, για τις χορηγήσεις. Βλέπετε δύο γραμμές. Το μπλε δείχνει την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Και έχουμε ξεπεράσει τις 25.000, αλλά βλέπετε και την κόκκινη γραμμή η οποία δείχνει το μηνιαίο επίδομα που έχει κατέβει πια στα 204 στη Γερμανία είναι πολύ λιγότερο από ό,τι ήταν στην αρχή του προγράμματος, αυτού που ήταν σχεδόν 300. Αν θέλαμε να έχουμε 300 και όχι 200 ευρώ, αυτό θα σήμαινε 15 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω το χρόνο, δηλαδή 50% περίπου. Έρχομαι τώρα στην πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση τη Κομισιόν από την οπτική γωνία των πανεπιστημίων έχει πολλέ ενδιαφέρουσε ιδέε. Καταρχήν, αύξηση του προπολογισμού. φυσικά. Απλοποίηση τη διαχείριση του προγράμματο, βεβαίω. Ενσωμάτωση των διεθνών προγραμμάτων τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Επίση, το να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα και σε επίπεδο μάστε με δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί όχι και επίσης ενίσχυση της συνεργασίας των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο το οποίο ενισχύεται με την πρόταση της Κομισιόν. Αλλά, αλλά, έρχομαι τώρα σε κάτι το οποίο με ενισχύει γιατί υπάρχει μια συστημική αλλαγή στο πρόγραμμα αυτό σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια. Με την ενσωμάτωση όλων αυτών των προγραμμάτων από το σχολείο μέχρι την διαβίου ε, εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ενηλίκων, η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο όμως εγκαταλείπει τα μεμονωμένα προγράμματα, ακόμα και προγράμματα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους. Και στη θέση όλων αυτών των προγραμμάτων τα οποία καταργούν και τα οποία είχαν μια κατανομή ανατομής, θα υπάρξει μια κατανομή κατατομής δράσης. Η δική μου πεποίθηση είναι ότι χρειαζόμαστε να κρατήσουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε τομέα και τα προγράμματα αυτά. Σας το λέω εδώ το γράφημα αυτό. Βλέπετε τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία θα περάσουν στο νέο σύστημα. Αυτά που είναι με κόκκινα γράμματα είναι αυτά που έχουν να κάνουν με το Πανεπιστήμιο και βλέπετε από την άλλη μεριά το Εράσμους για όλους που έχει ουσιαστικά μοναχά τρεις δράσεις. Στην ε, αριστερή πλευρά έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα όπου υπάρχει μια σαφής κατανομή και ταξινόμηση κατατομής. Δεξιά έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε ουσιαστικά ένα ανακάτωμα κατά κάποιο τρόπο ε, αμνών και ερυφίων ή μήλων και αχλαδίων. Για την πρόταση της Κομισιόν ακόμα περισσότερο. Το θέμα του ονόματος. Δεν θέλω τώρα να εμπλακώ στο θέμα αυτό. Το έρασμος είναι μια ακροστιχίδα είναι Ευρωπαϊκή Κοινοτική Δράση Κινητικότητας για τους Φοιτητές. Και το ερώτημα είναι αν ο Εράσμος πράγματι μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλους. Μήπως, μήπως γεννούμε προσδοκίες οι οποίες θα, θα μείνουν ανικανοποιητές στο τέλος. Αν δει κανείς τον προϋπολογισμό σε διάφορους τομείς, σίγουρα δεν μπορεί ο Έρασμος να καλύψει τις ανάγκες όλων, ιδίως η διεθνής του διάσταση οι προπολογισμοί για συγκεκριμένε δράσει και τομεί. Εντάξει, για τι δράσει έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η χρηματοδότηση κατά τομεί. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια σταθερότητα στον προπολογισμό και μια δυνατότητα σχεδίαση είναι απαραίτητη για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια και τη σταθερότητα στο σχεδιασμό. Και θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτή η σταθερότητα και στο πρόγραμμα. Το θέμα της απλοποίηση. ναι, αλλά θα πρέπει να ισχύει για όλους αυτούς. Η δίκηση δεν είναι μονάχα η διαχείριση χρημάτων και τεχνικών προδιαγραφών. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, περιλαμβάνει και το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων και κατά τη δική μας άποψη η ευθύνη για τα αποκεντρωμένα αυτά ε, διαχειριζόμενα προγράμματα θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών. Τέταρτον, η περιγραφή των προγραμμάτων όπως ελέγχθη προηγουμένως, είναι πάρα πολύ γενικόλογη και ασαφής. Είναι πολλά λεπτομεριακά στοιχεία τα οποία δεν τα ξέρουμε ακόμα. Ελπίζω ότι το πρόγραμμα θα είναι μάλλον καλύτερο από την περιγραφή που έχει δοθεί μέχρι στιγμής. Τα πανεπιστήμια έχουν αισιοδοξία σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, γιατί θεωρούν ότι με την συνένωση των ενδοευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο θα ενισχυθεί το πρόγραμμα. Επίσης, η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού σίγουρα θα λάβει υπόψη επαρκώς και τις ανάγκες της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης, το γεγονός ότι δίδεται έμφαση στην κινητικότητα πιστεύω ότι θα μπορέσουν και άλλοι τομείς να υποφελθούν από τρεις αυτές οριζόντιες δράσεις. Ελπίζουμε λοιπόν θα υπάρξουν πολλοί τομείς στου οποίου θα έχει επίπτωση το πρόγραμμα αυτό για τα άτομα, για την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά επίση και για μια μεγαλύτερη ελκυστικότητα στο διεθνή στίβο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Αυτό έχει να κάνει με καλύτερη συνεργασία. Θα θέλαμε όμως να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει δημιουργία ικανότητος και σε άλλα τμήματα του κόσμου, ιδίως στις εταιρικέ για μας περιοχές και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι σημαντικό λοιπόν και ο πολιτικός διάλογος, ο διάλογος για τις πολιτικές, συγγνώμη, με την διαδικασία της Μπολόνια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η συνεργασία με χώρες όπως τις χώρες της Ασίας θα πρέπει να ενισχυθεί και εξάλλου θα πρέπει να έχουμε και γέφυρες με άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως είναι η διαβιοεκπαίδευση. Έχουμε τώρα σε ορισμένε δράσεις του νέου προγράμματος που προβλέπονται όπως παρουσιάζονται στην πρόταση της Κομισιόν το σημαντικό μήνυμα το οποίο πρέπει να κατανοήσει ο πανεπιστημιακός χώρος είναι ότι όλες οι, όλα τα μέτρα τα οποία ισχύουν για τον πανεπιστημιακό χώρο θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και προστίθεται τώρα η νέα ε, στρατηγική προσέγγιση που έχει να κάνει με μια στρατηγική εταιρική σχέση. Αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Κατά δεύτερο λόγο, ε, δεν έχουμε μοναχά τα υπάρχοντα εργαλεία όπως είναι και η κινητικότητα στην Ευρώπη, αλλά έχει προσθεθεί και η διεθνής διάσταση, η οποία με την συνένωση του Εράσμους και του Εράσμους Μούντους έχει προκύψει και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Μπορεί κανείς να διαφυσβητήσει αν το ε, Εράσμους Μούντους θα πρέπει να πάψει να υπάρχει. Υπάρχουν πολλοί που το διαμφισβητούν αλλά είναι σίγουρο ότι πρέπει να υπάρχει μια διάσταση του προγράμματος Εράσμους και εκτός της Ευρώπης. Έρχομαι τώρα σε ένα τομέα ο οποίος προκύπτει από την ενσωμάτωση του Εράσμους Μούντους στο νέο πρόγραμμα και όπου υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και αφιβολίες. Εκεί που υπήρχαν στο παρελθόν κοινά προγράμματα μάστες και κοινά προγράμματα διδακτορικά, αυτό δεν θα υπάρξει πλέον. Για μένα είναι σφάλμα αυτό το γεγονός ότι αυτό μετακινείται στον, στη δράση Marie Curie. Μπορεί να φαίνεται από πολιτική άποψη ότι είναι μια καλή ενέργεια, αλλά ο τρίτος κύκλος, ο, ο κύκλος του διδακτορικού, που είναι το, ο τρίτος κύκλος στο σύστημα της Μπολόνια, ήταν ένα στοιχείο ελκυστικότητας μέσα στο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Και αν σπάσουμε τώρα με τα νέα αυτά μέτρα την διάσταση αυτή θα χάσουμε σε ελκυστικότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε αν θέλουμε πράγματι να ενσωματώσουμε την, ε, τα διδακτορικά μέσα στο πρόγραμμα Marie Curie. Επίσης, θεωρώ ότι η δυνατότητα να υπάρχει εγγύηση δανείων και αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εάν είναι συμπληρωματικό και όχι αντικατάσταση των προηγουμένων χρηματοδοτήσεων. Ένας άλλος τομέας όπου <clears throat> έχω κάποιες ανησυχίες είναι και η ενσωμάτωση του Tempus Α και του EduLink. Αναφέρθηκε ότι τα προγράμματα αυτά θα μπουν στην λεγόμενη διεθνή δημιουργία, διεθνούς χαρακτήρα δημιουργία ικανοτήτων με μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές οι οποίες είναι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αλλά θα θέλαμε να υπάρξει μια σαφ... μεγαλύτερη σαφήνεια για ορισμένες περιοχές όπως είναι η Κεντρική Ασία. Για το Α και για το Edge Link θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής είχαμε επικέντρωση στη Λατινική Αμερική και την Αφρική και εδώ το ερώτημα είναι πού θα τεθεί η Ασία, γιατί η Ασία είναι μια πολύ σημαντική Ήπειρος η οποία έχει ζωτικό χαρακτήρα για την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να μην λησμονηθεί η Ασία μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Κάποιοι άλλοι φόβοι οι οποίοι έχουν διατυπωθεί στον πανεπιστημιακό χώρο και οι οποίες διατυπώνται εδώ σε ερωτήσεις. Χάνουμε την ορατότητά μας και τη λεγόμενη sense of ownership, δηλαδή την ευθύνη που αναλαμβάνουμε για αυτά τα προγράμματα. Δεύτερον, η αλλαγή από μια προσέγγιση κατατομής σε μια προσέγγιση καταδράσης σημαίνει ότι έχουμε και μεγαλύτερη εστίαση σε μια πιο διοικητική προσέγγιση στο πρόγραμμα αυτό. Είναι κάτι που γίνεται μονάχα με στόχο τη διοικητική απλοποίηση. Δηλαδή, τρίτον, θα πρέπει να ανταγωνιστούμε για την απόκτηση κονδυλίων με άλλους τομείς εκπαιδεύσεως. Ελπίζω όχι και ελπίζω ότι η Κομισιόν το έχει κατανοήσει αυτό. Και τέταρτον, τι θα γίνει σε σχέση με την σταθερότητα στη χρηματοδότηση και τη δυνατότητα μακροχρόνιας στρατηγικής και πώς θα μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία χάραξη κατευθύνσεων. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με κατατομής προϋπολογισμούς. Κατά την δική μου άποψη <clears throat> θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία σε ένα συνδυασμό των τριών οριζόντιων γραμμών της Κομισιόν να συνδυαστούν με την ιδιαιτερότητα των τομέων μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι καμία αντίφαση στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά είναι μια, κατά την άποψή μου, θετική συμπλήρωση. Έρχομαι τώρα στα συμπεράσματα και στις συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να ενισχύσει την εκπαίδευση στην Ευρώπη και ίντραμούρος και εξτραμούρος και στο εσωτερικό της Ευρώπης και εκτός και θα πρέπει όχι μόνο να εξυπηρετήσει την Ευρώπη 2020 αλλά και τους στόχους της διαδικασίας του Μπολόνι. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αύξηση στον προπολογισμό ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις ε, δράσεις οι οποίες έχουν αποδείξει την αξία στο παρελθόν, να προσθέσουμε νέα στοιχεία και να διευρύνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την γεωγραφική εμβέλεια του προγράμματος αυτού. Πρέπει να δώσουμε καλύτερη επίσης πρόσβαση στο πρόγραμμα με καλύτερες υποτροφίες, με αντιμετώπιση ατόμων με ειδικέ ανάγκες για να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Τρίτον, θα πρέπει να κρατήσουμε τις προτινόμενες γραμμές δράσης, αλλά μέσα σε αυτές τις τρεις δράσεις θα πρέπει να έχουμε ειδικά, ειδικές υποδιαιρέσεις κατά τομής και να κρατήσουμε τα ονόματα για τις μέχρι στιγμής για του μέχρι στιγμή τομεί. Τέταρτον, να υπάρχουν σαφεί ελάχιστοι προπολογισμοί για του διάφορου εκπαιδευτικού στόχου και 80 με 85% του προπολογισμού θα πρέπει να είναι σταθερό για αυτά τα προγράμματα ω ελάχιστο επίπεδο. Τέλο, το πρόγραμμα πρέπει να είναι απλό, διάφανο και φιλικό προ το χρήστη και οι επιμέρους αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τις αποκεντρωμένες αρχές των κρατών μελών. Επομένως, Μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε την ήδη αρκετά ενδιαφέρουσα πρόταση της Κομισιόν και αυτό θα θέσει τα θεμέλια για μια νέα επιτυχή γενιά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δ. Βούτιχ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πάζη Ζάλβερ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτήν την συνάντηση σήμερα. Ε, ύστερα από τους τρεις προηγούμενους ομιλητές, εγώ θα παρουσιάσω την άποψη των μικρών χωρών του Βορρά. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα βρίσκομαι εδώ για να εξετάσω την πρόταση ε, προγράμματος μέσα από τέσσερα διαφορετικά πρίσματα. Πρώτον, ως Γενικό Διευθυντή της ΣΥΜΟ, Κέντρο Διεθνούς Κινητικότητας και Συνεργασίας στο Ελσίνκι, υπό την αιγίδα του Φιλανδικού Υπουργείου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης το οποίο απασχολεί 130 άτομα. Το ΣΥΜΟ υλοποιεί όλα τα προγράμματα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κατάρτισης, ε, του πολιτισμού, της νεολαίας και της παιδείας. Και ε, έχει διάφορα εθνικά και σκανδιναβικά σχήματα χρηματοδότησης. Δεύτερον, σας μιλώ ως κάποιος που τις τελευταίες δεκαετίες συμμετέχω στις προσπάθειες διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης, ιδίως στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Ε, το έργο ε, Στο έργο μου έχω μάθει να κατανοώ την αξία της διεθνοποίησης, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα άτομα να ανταποκριθούν στις πολύπλοκες καταστάσεις του σύγχρονου κόσμου. Το έχω καταλάβει αυτό από την ακαδημαϊκή μου καριέρα και από την επαγγελματική μου ιδιότητα. Επίσης έχω εργαστεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, στον ΩΣΑ και μέσα από αυτή τη δουλειά έμαθα να εκτιμώ τις ευκαιρίες που έχουν οι Ευρωπαίοι επειδή ζουν σε αυτό το πλούσιο και παλόμενο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό και ιστορικό περιβάλλον θα υιοθετήσω μια συστηματική ε, οπτική, μια γενικότερη οπτική σε σχέση με τους προηγούμενους ομιλητές. Πράγματι, το ευρωπαϊκό μέλλον έγκυται στα χέρια των νέων, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και υπό την έννοια της ειρήνης, της ευτυχίας, της κοινωνικής συνοχής. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους τα επόμενα χρόνια. Ήδη πριν από 250 χρόνια ο Βέντιαμιν Φραγκλίνος είπε ότι το να επενδύει κανείς στη γνώση αποδίδει πάντα τον μεγαλύτερο τόκο, τον υψηλότερο τόκο. Νομίζω όμως ότι εδώ στην Ευρώπη πρέπει να πιστεύουμε ότι η επένδυση στον άνθρωπο είναι η καλύτερη μακροχρόνια επένδυση. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε το νέο προτινόμενο πρόγραμμα το Erasmus for All, ο Erasmus για όλους, όπως είναι ο τωρινός του τίτλος. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι φυσικά ότι κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί ο κόσμος τα επόμενα 7 χρόνια και πώς θα επηρεάσουν οι εξελίξεις οι παγκόσμιες στην Ευρώπη. Κάτι που θα δούμε, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο είναι νέοι άνθρωποι που θα αναζητούν εργασία, σε, στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για, λίγους από αυτούς τους, για κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Όλο και περισσότερο τα έθνη μας γυράσκουν θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερος αριθμός ηλικιωμένων πολιτών ε, που θα είναι πιο εύποροι, πιο καλλιεργημένοι, πιο μορφωμένοι από τι προηγούμενες γενιές. Ε, επίσης, η κινητικότητα των ανθρώπων προσθέτει στην πολυμορφία της Ευρώπης, αλλά αυξάνει και τις πιθανότητες συγκρούσεων, ε, ακόμα και βίας. Όλες αυτές οι δυνάμεις πραγματικά θα συγκαθορίσουν πώς θα είναι η Ευρώπη και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό η Φινλανδία όπως και οι γειτονικές της σκανδιναβικές χώρες, έχει ωφεληθεί πάρα πολύ από τη συμμετοχή της στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20 χρόνια περίπου. Όταν μπήκε στο πρόγραμμα Έρασμος το 1992 η Φιλανδία, υπήρχαν περίπου 150 αλλοδαποί φοιτητέ που επέλεγαν την Φιλανδία ως τον χώρο των σπουδών τους στο, πλαίσιο των ανταλλαγών του εράσμου. Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι 6.000 ομάδες. Παρόμοιες τάσεις βλέπουμε και στα άλλα προγράμματα. Πράγματι, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπαιξαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την, ε, στην πρόθεση της διασυνοριακής κινητικότητας και συνεργασίας στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ο ένας στους δύο από τους εξερχόμενους και τα δύο τρίτα των εισερχόμενων φοιτητών χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus. Το πρόγραμμα Λεωνάρντο Νταβίντσι επίσης λειτουργεί και εκείνο και ευθύνεται για το ίμιση της διασυνοριακής επικοινωνίας και κινητικότητα στη Φιλανδία. Επίσης το ένα τρίτο των φοιτητών συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κομένιους. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για, την εκπαιδευτική, για τα εκπαιδευτικά ζητήματα στη χώρα μου. Η πρόταση που συζητούμε σήμερα εδώ αντιπροσωπεύει την συνέχεια των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η, πρόταση αυτή αναδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη σημασία που αποδίδεται στην νεολαία και στην εκπαίδευση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Η προτινόμενη αύξηση των πόρων είναι καλόδεκτη και απαραίτητη όμως για να επιτύχουμε τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα ωστόσο, Υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα στη σημερινή εκδοχή των προτάσεων. Επιτρέψτε μου να περιγράψω τα κυριότερα ζητήματα μέσα από το φιλανδικό πρίσμα. Γενικά υπάρχουν δύο τομείς ανησυχίας. Πρώτον, θα καλωσορίζαμε μια μεγαλύτερη έμφαση στη διαβίου μάθηση, με άλλα λόγια. Μεγαλύτερη επικέντρωση στη μεγάλη ιδέα του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον. Όπως το, είπε και Όπως το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ε, υπάρχουν άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας πεινασμένα για εργασία. Ο ρόλος της επαγγελματικής κατάρτισης ε, Ποιος είναι στην προαγωγή της εργασίας της απασχόλησης. Η σημερινή εκδοχή του προγράμματος αναγνωρίζει την ανάγκη αυτή. Δεύτερον, έχουμε ένα γυράσκοντα πληθυσμό στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Αυτό απαιτεί περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους ενήλικες. Από αυτή την άποψη η πρόταση σιωπά. Δεν λέει τίποτα για την ε, εκπαίδευση των ενηλίκων ή δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις ε, δυνατότητες ε, για, τον τομέα αυτό. Τρίτον, από τη στιγμή που τα σχολεία είναι οι μόνοι φορείς που καλύπτουν όλη την ηλικία, ε, τις, όλες τις κόρτες των μελλοντικών ε, Ευρωπαίων, θα πρέπει όλα τα σχολεία και οι σχολές να... Οι κοινέ ανάγκες όλων αυτών των ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, με συνέπεια. Ε, όλο και περισσότερο κινούνται ε, οι νέοι. Όλο και περισσότερες ε, κοινέ αξίες αναπτύσσονται, όλο και περισσότερες γέφυρες χτίζονται. Γι' αυτό θα πρέπει να διώσουμε περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας και κινητικότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο της σχολής ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος των υποψηφίων. Επίσης, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της νεολαίας απουσιάζουν από τη σημερινή πρόταση. Παράδειγμα, η κοινωνική ένταξη, η συμμετοχή των νέων, η ενεργός δράση, ε, ενεργός δράση τους ως πολίτες που είναι οι κύριες δυνάμεις των προγραμμάτων νεολαίας. Πιστεύουμε ότι η πρόταση μπορεί να βελτιωθεί εάν όλες αυτές οι εκφάνσεις τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Το μελλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει γενικά να είναι πιο ολιστικό και θα πρέπει να επιφέρει μια καλύτερη ισορροπία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαφορετικών ε, στοχευόμενων τομέων. Ο τομέας της νεολαίας, της νεότητας, θα πρέπει να του δοθεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και θα πρέπει να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο κονδύλιο για την εκπαίδευση ενηλίκων. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία όμως έχει η νέα, η νέα πρόταση κανονισμού να να δώσει κονδύλια και χρηματοδότηση σε όλες τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, να χρηματοδοτηθούν όλοι οι τομείς. Διαφορετικά, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταλήξουμε κάπου που δεν έχουμε ιδέα τι θα είναι. Δεύτερον, θα θέλαμε να δούμε συνεργασία με τρίτες χώρες, να ανοίξει αυτό για όλους. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, από τις εξωτερικές σχέσεις και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Γι' αυτό έχει ύψιστη σημασία όποτε γίνεται, όποτε αυτό είναι δυνατό, οι νέοι και οι ενήλικοι φοιτητέ να μπορούν να έρθουν σε επαφή και να συστήσουν φιλίε όχι μόνο εντό τη Ευρώπη, αλλά και έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να ιδωθεί ε, σε απομόνωση από τους γειτονές της και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ίσως να αποδειχθεί ε, κοντόφθαλμο ίσως φανεί κοντόφθαλμο ότι η συνεργασία με τις τρίτες και τις γειτονικές χώρες ε, περιορίζεται μόνο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ε, το πρόγραμμα εκτείνεται μέχρι το 2020. Είναι δύσκολο να φανταστούμε πώ θα είναι η Ευρώπη μέχρι τότε. Ίσως οι γείτονέ μα στη Βόρειο Αφρική να ωφεληθούν από τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά σχολεία επαγγελματική κατάρτιση, ή είδο τα σχολεία τη Ευρώπη, να καταστούν καλύτερα εάν τα δίκτυά τους ε, συμπεριλάβουν και ανατολ, ανατολικούς γειτονέ μα Στον τομέα τη ε, εν, εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάτι που μπορεί να συστήσει συνεργασίε με ολόκληρο τον κόσμο. Από το με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο τομέας της νεότητας έχει ε, διεξάγει διάφορες δράσεις και έχει ενισχύσει την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας των πολιτών, στις ε, ε, γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αλλού. Φοβούμεθα ότι η τωρινή κατανομή πόρων δεν θα επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Εδώ λοιπόν, ειδού λοιπόν η πρότασή μας. Ας αφήσουμε τις πρώτες ανοιχτές στο νέο πρόγραμμα για συνεργασία με τρίτες χώρες σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο στην νεότητα και στην ανώτατη εκπαίδευση. Ίσως απρόβλεπτες αλλαγές στην ε, στο γεωγραφικό μας χώρο να απαιτήσουν βαθύτερη και ευρύτερη συνεργασία εκτός των συνόρων μας. Κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτά τα θέματα, αυτές τις πηγές ανησυχίας, θα ήθελα να εξετάσω την πρόταση υπό το πρίσμα ε, των κρατών μελών. Αυτή η πρόταση του Erasmus for All τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία του πρέπει να εξεταστούν με προσοχή. Να πω κάποια στοιχεία. Πρώτον, θεωρούμε ότι η πρόταση ε, ορθολογικοποίησης και ομογενοποίησης είναι θετική. Η πείρα έχει δείξει ότι τα σημερινά προγράμματα έχουν πάρα πολλές μορφές δράσεων, συχνά πολύ μικρές, περιορισμένες, μικρής κλίμακας και δεν μπορούν να έχουν ε, πραγματικό αντίκτυπο. Τα πανεπιστήμια έχουν διαφορετικές ανάγκες από τις ομάδες νεότητας Ωστόσο, πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρο εξορθολογήκευση. Μπορούμε να δούμε πώ το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί. Η απλοποίηση θα είναι ευεργετική για τους πελάτες και θα αυξήσει την ε, αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και στη διοίκηση, πράγμα απαραίτητο στη σημερινή οικονομική κατάσταση. Η αποκέντρωση δημιουργεί καλύτερο αντίκτυπο και λιγότερο διοικητικό βάρος. Τα προγράμματα νεότητας και εκπαίδευσης όταν είχαν πρωτοδημιουργηθεί στα τέλη δεκαετίας του 90 τότε η διαχείριση των προγραμμάτων ήταν συγκεντρωτική εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, με τα χρόνια αυτό έχει αλλάξει καθώς η επιλογή των προγραμμάτων ε, αλλά και η διαχείριση έχει ανατεθεί σε εθνικούς φορείς και στις συμμετέχουσες χώρες επίσης. Η άνοδος, της, αυξημένη αποκέντρωση των έργων και των, της διαχείρισης των προγραμμάτων υπήρξε αναντήρητη επιτυχία των ε, υφιστάμενων προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά έγιναν για το λόγο αυτό πιο προσβάσιμα προς τις ομάδες στόχους και, έχουν, και βελτίωσαν την αποτελεσματικότητά τους. Αυτή η τάση ασφαλώς θα πρέπει να συνεχιστεί. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας ωστόσο δεν είναι σαφής ως προς αυτό και θα πρέπει πιστεύω να εξειδικευθεί περαιτέρω έχει ζωτική σημασία επιπροσθέτως των δράσεων στρα... κινητικότητας να να αποκεντρωθεί και η σύναψη στρατηγικών συμπράξεων. Η εθνική συνιστόσα, πιστεύω, αυξάνει την ε, συνέπεια, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα. Στην Φιλανδία η διαχείριση ανήκει στην ε, ΣΥΜΟ, τον Εθνικό Φορέα της Φιλανδίας. Ε, ο Σίμος, η αρχή αυτή η φιλανδική συχνά ε, αναφέρεται ως ε, πρότυπη, ως καλό παράδειγμα. Καλό είναι ένας φορέας ε, να, έχει, να συγκεντρώνει σε αυτές τις αρμοδιότητες, ιδίως για χώρες που έχουν το ίδιο μέγεθος με την Φιλανδία. Ε, στην Φιλανδία έχει αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η κινητικότητα, η συνεργασία, αλλά και ο αντίκτυπος, ε, ε, η επίδοση ήταν καλύτερη και αυτό αναγνωρίστηκε από όλους. Σημασία έχει επίσης η Εθνική Φορή Υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να έχουν στη διάθεσή τους χρόνο και πόρους πέρα από την, ε, που να καλύπτουν κάτι πέρα από την καθημερινή τους εργασία. Ε, ασφαλώς θα πρέπει να ανοίξει ο εγχώριος διάλογος για τη διεθνοποίηση των κοινωνιών μας. Επιπλέον, αναπτύσσουμε και νέους τρόπους αξιολόγησης του αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων ε, δραστηριοτήτων ευρωπαϊκών συνεργασίας. Σύντομα, θα θέσουμε σε εφαρμογή πιλωτικές εφαρμογές για να δούμε πώς μπορούν οι νέοι να αποκτήσουν σφαιρική παγκόσμια οπτική ε, με τρόπο που να ενισχύει τις αξίες αλλά και την ευεξία τους κατά συνέπεια της συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα συμπεριλαμβάνουν εκείνο που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποδείξει την αξία τους και τη συνεισφορά τους στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στον τομέα της νεότητας και για τις κοινωνίες μας ε, κατ' επέκταση. Βελτιώνουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν ε, όσους ε, έχουν λιγότερες ευκαιρίες σε σχέση με άλλους τα προγράμματα αυτά είναι από μεταξύ των λίγων εργαλείων που είναι άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες της Ευρώπης. Η συμμετοχή στα προγράμματα ε, ε, ενισχύει μια νέα γενιά, η οποία είναι πιο ανοιχτή στις διαφορετικές κουλτούρες, έχει μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος και είναι λιγότερο ξενόφοβη. Ε, υπηρετείται έτσι το ευρωπαϊκό ιδανικό για την κοινωνία. Πιστεύω ότι τα εργαλεία αυτά θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο και στη Φουλανδία αλλά και στις υπόλοιπες ε, χώρες μέλη, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση και ενισχύοντας το ευεξία των κοινωνιών μας. Η σκανδιναβική οπτική είναι πολύ ιδιόμορφη λόγω της γεωγραφίας των χωρών αυτών αλλά και λόγω της σημασίας της διεθνοποίησης στις βόρειες αυτές χώρες. Εάν θέλουμε να κάνουμε έξυπνη χρήση των, του σχετικά μικρού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος καλύτερος τομέας από την επένδυση στους ανθρώπους, στην παιδεία, στο κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος είχαμε ένα ευρύ φάσμα απόψεων, επένων, επικρίσεων για την πρόταση της Κομισιόν. Δόξα το Γιαραμπή, ακούσαμε και στο τέλος την, ε, ακούσαμε ενδείξεις ότι πράγματι ελήφθησαν υπόψεις και οι απόψεις της κοινωνίας θα ήταν χρήσιμο να είχαμε καλέσει και ένα ευρύτερο ε, αριθμό ομιλητών αν αυτό ήταν δυνατό. Εμείς πάντως θα πρέπει να δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια ποια θα είναι η στάση μας. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τους συναδέλφους να δείξουν αυτοσυγκράτηση στις παρεμβάσεις τους για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Η κυρία Νεβεντέλοβα από τη Σλοβακία έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες ε, για τις λεπτομερείς εξηγήσεις που μας έδωσαν σε ό,τι αφορά τις θέσεις τους. Ίσως κάποια στοιχεία να χάθηκαν βέβαια στην πορεία. σε ό,τι αφορά τι συγκεκριμένε σα προτάσεις για το Erasmus for Τι αλλάζετε λοιπόν κύριε Μάτσης στην ε, τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής. Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξουν ε, οι προτεραιότητε, ο τίτλο, Ποια είναι τα πρακτικά, τα στοιχεία που μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεύτερον, θεωρείτε ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης ε, ε, αντικατοπτρίζεται επαρκώς μέσα στην πρόταση της Επιτροπής. Εμείς ε, δεν θεωρούμε ότι καλύπτονται και προσωπεύονται όλες οι ομάδες ηλικιακές επαρκώς. θεωρείτε λοιπόν επαρκές το πρόγραμμα της Επιτροπής. Πιστεύετε ότι θα ωφελήσει όλο ένα και περισσότερους νέους να έχουν πρόσβαση στην, ε, στην κατάρτιση κατά την Επιτροπή αυτό είναι φυκτό. Εσείς συμφωνείτε? Τάκουλα. Μερσή λέει πρόεδρος. Κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα, να θέσω πολλά ερωτήματα καταρχήν για το πρόγραμμα αυτό. Ας μιλήσουμε όμως λιγάκι για τον προϋπολογισμό του λέτε ότι θα αυξηθεί ο προπολογισμό, αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Γιατί φυσικά η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πρέπει να τονίσουμε ότι τα προγράμματα αυτά γίνονται για τους ανθρώπους και όχι για τους διοικητικούς. γι' αυτό, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Βούτιχ, πραγματικά αναρωτιέμαι αν υπήρξε κάποια μετατόπιση παραδείγματος σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν περάσαμε από προγράμματα μεμονωμένα κατά τομής σε ένα πάρα πολύ άμορφο λιγάκι πρόγραμμα και μια πιο πλήρη αντιμετώπιση. Περάσαμε ουσιαστικά από μικρομάγαζα σε ένα είδος εμπορικού κέντρου. Δεν ξέρω αν τα βλέπω σωστά αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ανάγκη της ε, διαβίου εκπαίδευσης, ελπίζω ότι το να βρίσκεται σε ένα εμπορικό κέντρο επιτρέπει στον καθένα να βρει το μαγαζί το οποίο τον ενδιαφέρει. Ελπίζω λοιπόν ότι τόσο οι νέοι όσο και οι πιο ηλικιωμένοι, εφόσον ο πληθυσμός μας γυράσχει σταθερά, θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν την κατάλληλη εκπαίδευση και αυτή που είναι πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Βλέπω λοιπόν να υπάρχει αυτή η αλλαγή παραδείγματο από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ίσως όλα αυτά θα πρέπει να μα οδηγήσουν στο να σκεφτούμε λίγο περισσότερο γιατί τονίζω ότι για μένα το πρόγραμμα αυτό δεν είναι για του διαχειριστέ, αλλά για του ε, τελικούς αποδέκτες, για τα άτομα. Για το Κομένιους. Το Κομένιους ήταν πράγματι μια ιστορία επιτυχίας. Γνωρίζουμε τις μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι το Κομένιους δεν προσέφερε πραγματικά σε επίπεδο προσθέμενης αξίας στην Ευρώπη. Σε τελική ανάλυση δεν παρέχει προσθέμενη αξία, απλώς δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να ταξιδεύουν δεξιά και αριστερά και να έχουμε ανταλλαγές, αλλά αυτό δεν έχει οδηγήσει σε προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω λοιπόν αν και το Κομένιους θα έπρεπε να υποστεί κάποιες αλλαγές σε σχέση με τις πρακτικές του. Και ένα ακόμα ερώτημα που θέλω να θέσω. Θεωρείτε να υπάρξουν και αλλαγές ε, στο Κομένιους για να περιλαμβάνει και το, το δημοτικό και να υπάρξει και εκεί κάποια προσθέμενη αξία. Θα σας δώσω ότι, να πάτε στη δική μου, λέει η κυρία Πάκα, αλλά δεν είμαι δυστυχώς εμπειρογνώμων. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμενους για τις παρουσιάσεις τους. Ως Φιλανδός, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Κάποιος αναφέρθηκε στο νέο μέσο εχεγγύων για τα δάνεια. Πράγματι, στην, στο πρόγραμμα της Μπολόνια συμφωνήθηκε ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπίσει το δικό του σύστημα δανείων για τους ε, φοιτητές. Τώρα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ίσα. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου υπάρχουν τέτοια συστήματα ε, διασφάλισης των φοιτητικών δανείων. Και τώρα το θέμα είναι αν είναι αρκετά ελκυστικά αυτά τα δάνεια και τα συστήματα για τους φοιτητέ. Και ακούω ότι ορισμένες ομάδες ε, δεν επιθυμούν αυτά τα συστήματα. Κάποιος ανέφερε ότι πολλοί από αυτούς τους φοιτητές ε, τελικά καταλήγουν άνεργοι και εκεί είναι ιδιαίτερα δύσκολο το να αναλάβει κάποιο και ένα δάνειο. Ιδιαίτερο εν μέσω μιας κρίσης χρέους. Εξάλλου, δεν θέλουν όλες οι τράπεζες να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα. Επομένω, πώς είναι δυνατόν να έχει κάποιος πρόσβαση, κάποιος, ε, να έχει κάποιος πρόσβαση σε ένα τέτοιο δάνειο σε άλλο κράτος μέλος η Επιτροπή πώς θα διασκεδάσει αυτούς τους φόβους. Ουσιαστικά θέλω να πω ότι ο κόσμος φοβάται. Φοβάται ότι αυτά τα προγράμματα που μπορεί να μην συνεχιστούν και τότε τι ακριβώ θα κάνει η Επιτροπή και για την επαγγελματική κατάρτιση και για την επίσημη εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχει αντιμετωπίσει η Κομισιόν και ίσως εκεί <clears throat> υπήρξε κάποια παρεξήγηση για αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν. κυρία Κώστα τώρα. Θα ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ στους εμπειρογνώμονες γιατί με μεγάλη ποιότητα συνέβαλαν και με μεγάλη σαφήνεια. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, αν υπάρχει συνοχή μεταξύ των παρεμβάσεών τους. Ε, παρόλο που πραγματικά είναι σημαντικό να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, ε, με περισσότερα κονδύλια, όλοι τα είπαν αυτά ωστόσο διατύπωσαν και κάποιες επικρίσεις που είναι σημαντικές. Είναι σημαντικό νομίζω να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Θα κάνω ερωτήσεις στους δύο εμπειρογνώμονες πάνω σε τρία ε, σημεία. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η Επιτροπή το όνομα του προγράμματος, ο τίτλος, είναι κάτι πολύ αποτελεσματικό γιατί είναι, έχει έναν επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά το περιεχόμενο είναι ακόμα σημαντικότερο κατ' με. Το Youth Forum, ε, δύο ερωτήσεις για το Youth Forum. Από τι κατάλαβα, θέλουν, αποδίδουν μία αυτονομία στο πρόγραμμα Youth in Action, ζητούν μάλλον μια αυτονομία. Ε, ε, και αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορούν να το συνδυάσουν με τον αθλητισμό. Πρώτο ερώτημα για τα Masters. Ε, υπάρχει κάτι θετικό στην πρόταση αυτή. Είναι μια νέα ευκαιρία που προστίθεται από ό,τι κατάλαβα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις υποτροφίες, αλλά θα υπάρξει ένα ταμείο εγγυήσεων το οποίο θα βοηθήσει τους φοιτητές που δεν μπορούν αλλιώς να κάνουν ένα Master. Το Youth Forum τι άποψη έχει γι' αυτό και υπάρχει έχει κάποια πρόταση να διατυπώσει. Ε, στη δική μου χώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλουν να υπάρξει ένα μεικτό σύστημα και υποτροφής και πρόσβαση στις, στο Ταμείο αυτό των εγγύησεων δανείων. Εγώ συμμερίζομαι τα θέματα που έθιξαν οι εμπειρογνώμονες ε, πάνω στην διαβίου μάθηση προοπτικά, ιδίως στο πρόγραμμα Κομένιους, το οποίο ειδικά απευθύνεται στις σχολές. Και αναρωτιέμαι, τα οι στοχευμένες σχολές συγχέονται με τις υπόλοιπες ε, αυτό το μείγμα που προτείνει ο κύριος Βούτιχ, αν δεν κάνω λάθος, ε, στο τέλος. Το μείγμα μεταξύ δράσεων και τομέων που νομίζω πως είναι μια προσέγγιση που θα μπορούσε πραγματικά να συνενώσει τόσο τις οριζόντιες δράσεις και χωρίς να χάνει από τα μάτια τις ε, διαχωριστικές γραμμές επίσης μια απλοποίηση, μια απλοποίηση στη διαχείριση. Υπάρχει όμως ε, ένας κίνδυνος να υπάρξει μια σύγχυση ως προς τους στόχους, να μην διακρίνουμε μεταξύ των διαφορετικών στόχων. Το να υπάρχουν διαφορετικοί διακριτοί στόχοι είναι ένα μακροπρόθεσμο θετικό στοιχείο. Ε, είναι διαφο... Ε, πολύ δύσκολο να οικοδομηθεί ένας, ε, ένα κεκτημένο, ένα σώμα γνώσεων χωρίς αυτές τις διακρίσεις. Πάρα πολλοί εμπειρογνώμονες ε, από πολλές χώρες έχουν θέσει το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι έχουν γίνει ακουστοί. Σας ευχαριστώ. Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες οι οποίες κάνανε μια πολύ, κάνανε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και μας ε, έχουν δώσει πολλές πληροφορίες. Θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο που εκφράζει και τις δικές μου προσδοκίες ότι παραδείγματο χάρη το καινούριο κεφάλαιο συμμετοχή των νέων στον έρασμο ή άλλα κεφάλαια θα μπορέσουν να παραμείνουν συμβατά με αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα ως προγράμματα. Να σας δώσω το παράδειγμα της Αυστρίας. Υπάρχει μία ε, ένωση νέων που καλύπτει όλο το έδαφος της Αυστρίας. Υπάρχει ήδη μία δομή η οποία είναι έτοιμη και λειτουργεί και η οποία πρέπει να παραμείνει μέσα στο πλαίσιό της. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί η υπόψη ημέρημνα να παραμείνουν οι δομές αυτές. Επίσης τώρα στέκομαι στο σημείο της ε, ε, κινητικότητας ότι αυτό φυσικά θα πρέπει να έχει μεγάλη προτεραιότητα αλλά η στοχοθεσία θα πρέπει να κινείται γύρω από την Ευρώπη 20 και 20. Όχι μονάχα γύρω από την κινητικότητα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κινητικότητα. Ή η αύξηση του ποσοστού φοιτητών στα πανεπιστήμια. Και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα με την κινητικότητα. Επίσης είναι απαραίτητο αυτές οι έννοιες αυτά τα προγράμματα να εξυπηρετήσουν τις απόψεις αυτές που ανέφερε ο πρόεδρος Μπαρόσο πρόσφατα στη Βιέννη ως βασικά στοιχεία benchmarking για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Η δυτή δηλαδή μορφή της εκπαίδευσης και κατάρτισης εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη σαφήνεια κατά την απόψή μου. Χωρίς, χωρίς μικρόφωνο, κύριος Πιτέλλα. Πρόεδρε, θυμάμαι με περηφάνεια ότι παρουσία τη δική σας και άλλων συναδέλφων υπήρξαμε μεταξύ των ε, υπέρμαχων της διεύρυνσης της εκπαίδευσης και αλλού. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι οι ε, νέοι μας μεγαλώνουν σε μια κοινωνία εντελώς διαφορετική από αυτή που γνώρισαν οι γονείς τους. Υπάρχει η τεχνολογία της πληροφορικής και όλες οι άλλες αλλαγές που έχουν υπησέλθει. Πώς, μπορούμε να έχουμε μια πιο στενή διασύνδεση μεταξύ των προγραμμάτων για τους νέους και των νέων μέσων ε, περιφερειακής πολιτικής. Πώς θα, κάνουμε τη διασύνδεση με τη συμμετοχή σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την εκπαίδευση των νέων και το πρόγραμμα Εράσμους όπως και το Κομένιους. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα προγράμματα όχι μόνο για την παιδεία των νέων αλλά για να μπορέσουν οι νέοι να προσεγγίσουν καλύτερα τη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό έχουν την εμπειρία της πρόοδου που έχει επέλθει με την ε, ευρωπαϊκή πορεία. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τους εμπειρογνώμονες ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την ανάγκη να βελτιωθεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών η γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών. Εγώ πάντα υποστηρίζω κάτι τέτοιο και αυτό φαίνεται και από εκθέσεις της Επιτροπής μας, η έκθεση Lockhart, η έκθεση Καβαντά πέρσι που αναφέρεται στο σημείο αυτό, ότι είναι απαραίτητο να ενσωμετωθούν στα ε, εκπαιδευτικά προγράμματα, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο πρώτου κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών, μαθήματα σε σχέση με τους θεσμούς και την ιστορία της Ευρώπης για να γνωρίζουν καλύτερα οι νέοι την ιστορία, τους στόχους και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και έτσι να μην υπάρξει αυτή η απόσταση <clears throat> που οδηγεί πολλέ φορέ σε αδιαφορία των νέων σε σχέση με την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόρις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, των οργανώσεων νέων. Έχουμε λάβει εκατοντάδες email και ερχόμαστε σε επαφή με πολλές από αυτές τις οργανώσεις ε, στις περιφερειές μας, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις αλλαγές ε, στις οργανώσεις νέων και στα σχολεία και στις οικογένειες. Βεβαίως, θα πρέπει να απαντήσουμε το εξή ερώτημα γιατί αλλάζουμε αυτά τα συστήματα. Νομίζω ότι οι στόχοι του ορίζοντα 2020 είναι ξεκάθαροι. Όλοι βλέπουμε τα δημογραφικά προβλήματα. Ξέρουμε ότι έχουμε τεράστιο ζήτημα με τις ε, ε, δεξιότητες ε, των Ευρωπαίων. Βλέπουμε ότι τα σχολεία, τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς των αλλαγών που έχουν επέλθει και λόγω κρίσης και λόγω εξελίξεων ε, στην τεχνολογία. Υπάρχει όμως πρόβλημα με την ανεργία των νέων, γιατί δεν υπάρχουν πλέον εχέγγυα ούτε από τα σχολεία, ούτε από την αγορά εργασίας. Όμως Έχουμε ορισμένα πολύ καλά προγράμματα όπως το Εράσμου, το Κομένιους, πολύ καλά προγράμματα και υπάρχει το ερώτημα γιατί το, τα αλλάζουμε. Ε, αποδέχομαι το επιχείρημα της Επιτροπής για την προώθηση, ε, την ενσωμάτωση αυτών των προγραμμάτων για την απλοποίηση των διαδικασιών. Αλλά θα πρέπει να θέσουμε το εξή ερώτημα. Είναι καλύτερο να έχουμε αυτά τα προγράμματα ως ξεχωριστά ή να έχουμε ένα πρόγραμμα ναυαρχίδα ε, με ανεξάρτητα ε, προγράμματα στο ιστορικό του. Το, το πρόγραμμα Greenwich που είναι τόσο σημαντικό για τους ε, μεγαλύτερους ηλικία, το πρόγραμμα Leonardo ε, που βοηθά την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ανεπίσημη εκπαίδευση που ανέφερε ο εκπρόσωπος των νέων. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σα. Εγώ όμω θα ήθελα να έχουμε διασφαλίσεις ότι καθένα από αυτά τα προγράμματα θα είναι ανεξάρτητο και θα, έχουμε, θα υπάρχει και ε, γραμμή προπολογισμού. Αλλά θα υπάρχουν και χέγγια για την συνέχιση της δράσης και παρακολούθηση της δράσης. Τι πιστεύετε όμως εσείς. Oh, Κυρία Μεταγκρίζα, δεν ξέρω το όνομά σας. Ναι, ναι, πίσω από τον κύριο Πιτέλα. Προσπαθούμε να βρούμε τα ονόματά σας, αλλά δεν, τα βλέπω πια. Ονομάζομαι η Κώστελο, είμαι καινούρια ευρωβουλευτής από την Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, έχουν την δυνατότητα να μιλήσω εδώ σήμερα. Ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα, γιατί για δέκα χρόνια ήμουν διευθύντρια μιας εθνικής ε, Υπηρεσία ε, ενός εθνικού οργανισμού και έχω και εγώ κάποια εμπειρία. Δυστυχώ δεν πρόλαβα όλες τις, τις ε, ε, παρεμβάσεις γιατί ήμουνα στην Επιτροπή ΑΦΕΤ προηγουμένω. Άκουσα όμω κάποιες από τις παρεμβάσεις. Το πρώτο που θα θέλω να πω είναι ότι συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις κάποιων μελών για τον τίτλο του προγράμματος. Ε, και για το Εράσμους. Ε, γνωρίζω ότι έχουμε περάσει πολλά χρόνια για την οικοδόμηση του ε, ονόματος του Κομίνη, του Λεωνάρντο και όλα αυτά και δεν νομίζω ότι έχει, νόημα τώρα να, τα κάνουμε όλα αυτά Εράσμους και να τα προωθήσουμε όλα αυτά ως Εράσμους. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε κάποια συστήματα για την ενεργεία των νέων και είπαμε ότι έχουμε 7,5 εκατομμύρια ανέργους, ε, νέους ανέργους στην Ευρώπη. Συζητήσαμε κάποιες από τις λύσεις για αυτό το θέμα ε, και σε σχέση με κάποια από τα προγράμματα. Μία από τις λύσεις που αναφέρθηκαν είναι το ζήτημα της επαγγελματικής κατάρτισης και της έλλειψης αυτής και της έλλειψης ελκυστικότητα τη επαγγελματική κατάρτιση. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα μέλη που αναφέρθηκαν σήμερα αναφέρθηκαν στο Εράσμου και όχι στο Λεωνάρντο. Υπάρχει λοιπόν ε, μια σύγχυση για την, ε, για την προώθηση των προγραμμάτων, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μείνουν όσοι έχουν τα πράγματα και συμφωνώ με την διατήρηση των ξεχωριστών προγραμμάτων. Ναι, έχουμε λοιπόν διαφορετικό πρόγραμμα για τους νέους, για τον επίσημο και ανεπίσημο τομέα. Για τις άλλες ε, προτάσεις που αναφέρθηκαν, για την έλλειψη κινητικότητας, για τους ε, ενήλικες, πράγματι υπάρχει έλλειψη, έλλειψη κινητικότητας και αυτό είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα εδώ να μιλήσω. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσεί πώ μπορώ να, να, να συμβάλλω περαιτέρω και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Είμαστε στην αρχή, στα Σπάργανα. Η έκθεση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο και μετά μπορείτε σε όλες τις καλοκαιρινές σας διακοπές να σκέφτεστε για τροπολογίες. Ελπίζω ότι δεν θα είναι πάρα πολλές οι τροπολογίες βέβαια. Ο... Η κυρία Κάμα Εβερτ και μετά θα δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους ε, ομιλητές μας. Νομίζω ότι πάρα πολλά από αυτά τα οποία ακούσαμε συνδυάζονται με τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως το πρωί στην Επιτροπή μας. Είχα μονάχα ένα σύντομο ερώτημα στον εκπρόσωπο της νεολαίας. Είχαμε ξεκινήσει με την πανοκρουσία ουσιαστικά αυτή τη νέα στρατηγική για τους νέους πριν από ένα-δύο χρόνια. Και άμα κοιτάξει κανείς αυτό το πρόγραμμα, βλέπουμε ότι αυτή η στρατηγική για τους νέους δεν παίζει πια κανένα ρόλο. Κάτι το οποίο λιγάκι μας εκπλήσει. Δεν έχει νόημα να την βάλουμε ξαφνικά στο σιρτάρι και να την ξεχάσουμε. Έχετε κάποιες ε, ιδέες σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα για τους νέους, πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τα στοιχεία αυτού του προγράμματος με τη στρατηγική που διαγράφει τώρα η Κομισιόν. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε έναν τρόπο να συνδέσουμε αυτά. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Θα ήμουν ευγνώμων αν είχατε κάποια τέτοια πρόταση να κάνετε. Ωραία λέει η πρόεδρο. Και τώρα οι εμπειρογνώμονε θα λάβουν το λόγο. Μπορείτε να απαντήσετε με τη σειρά που θέλετε εσεί, Παρακαλώ κύριε Σπίγκελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω το ερώτημα που αφορά τα θέματα της ε, σχολικής εκπαίδευσης. Αν ε, πρόκειται να αλλάξω κάποια πράγματα στο πρόγραμμα, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τα ονόματα των τομέων, να κρατήσουμε τους τομείς και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με το πρόγραμμα, γιατί είναι πάρα πολύ ασαφές αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι έτσι απαντώ το πρώτο ερώτημα. Τώρα για την διαβίου εκπαίδευση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η επιτυχία αλλά και το κομμένιους. Δεν μπορεί κανείς πάντα να καταμετρήσει τι προκύπτει από την σχολική εκπαίδευση. Όταν έχετε τα παιδιά ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρουν από νεαρή ηλικία τι κάνει η Ευρώπη και πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κερδίσουν πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στις μεταγενέστερες σπουδέ τους και στην επαγγελματική ζωή τους. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ μια θεσμική προσέγγιση αν δούμε τι καταφέραμε με τη μετεκπαίδευση των ε, ε, διδασκόντων. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο αριθμό των ε, αιτήσεων θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πιο θετική αντιμετώπιση σε όλα αυτά με ένα θεσμικό χαρακτήρα για τα προγράμματα αυτά, για το Κομένιους. Πιστεύω, είπε κάποιος ότι έχουμε χάσει τη στοχοθεσία. Νομίζω ο Ιταλός συνάδελφος, η Ιταλίδα συνάδελφος νομίζω, χρειαζόμαστε κάποιους ε, τομείς που να καταλαβαίνουμε ποια είναι η στοχοθεσία. Νομίζω και το Κομένιος είναι ένα καλό πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοιχτό για τους αποδέκτες και όπου μπορούν και οι πολίτες να καταλάβουν τη σημασία του. Πάλι από κάποιο Ιταλό συνάδελφο, το θέμα των νέων μέσων ενημέρωσης, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι οι οποίοι μεγαλώνουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην εκπαίδευσή τους στα νέα μέσα ε, πληροφόρησης. Με την ε, ηλεκτρονική αδελφοποίηση πιστεύω και με τέτοιες συνεργασίες μπορούν να ενισχυθούν αυτές οι ενέργειες. Το ερώτημα του αν χρειαζόμαστε ένα ιδιαίτερο μάθημα για την Ευρώπη, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ε, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπερφορτώνουμε τα σχολεία με μαθήματα όπως η Ευρώπη, ένα μάθημα για την οικονομία, την ευρωπαϊκή κτλ. Ένα πράγμα είναι το να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αφηρημένα και άλλο είναι να λειτουργεί κανείς μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Τώρα για τις λεπτομέρειες τι κάνει η Κομισιόν και τι αρμοδιότητες έχει, όλα αυτά μπορεί να τα διαβάσει κανείς άμα χρειαστεί. Στο ερώτημα γιατί πρέπει να σταματήσουν ορισμένα προγράμματα που έχουν αποδείξει την αξία τους. Όχι, δεν θέλω να σταματήσουν. Πρέπει να διατηρηθούν. Ο κάθε τομέα, θα πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του. Και αυτό γίνεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση του προπολογισμού για κάθε τομέα. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε μια αξιοπιστία και μια συνέχεια και μια σταθερότητα και σε ό,τι αφορά τους εθνικούς φορείς. Υπάρχουν δομές που υπάρχουν ήδη. Αν υπάρξει απόλυτη ευκαμψία στον προπολογισμό, δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα κάνει γιατί δεν ξέρει πόσες αιτήσει θα έχει. Ε, εντάξει, αυτά. Εκπρόσωπος της νεολαίας ο κ. Μάτουσέκ. Ευχαριστώ πολύ για το πρώτο ζήτημα τη απλούστευση. Εμεί δεν είμαστε αντίθετοι. Πιστεύουμε ότι αυτό είπαν και οι νέοι μετά την αξιολόγηση. Ναι, θέλουμε τον εξορθολογισμό και όλα αυτά. Αλλά εξαρτάται για το τι εννοούμε με όλε αυτέ τι έννοιε. Θέλουμε ένα πιο εύκολο και πιο γρήγορο ε, πλαίσιο με ε, πιο διαφανείς διαδικασίες και, και ούτω καθεξής. Αν αυτό εννοείται με απλούστευση, συμφωνούμε προς το παρόν η πρόταση της Επιτροπής δεν ε, περιλαμβάνει τίποτα από αυτά που υπάρχουν σε έναν οδηγό χρήση αν θέλετε. Αλλά εσείς ως δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι των ε, Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να εκφέρεται γνώμη για το πώς θα πρέπει να ε, καταρτιστούν αυτοί οι κανόνες και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπόλογη με τη δημοκρατική έννοια. Γι' αυτό όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό, τουλάχιστον κάποια αναφορά, για να ξέρουμε ότι οι έννοιες για τις οποίες μιλάμε θα εγκρίνονται μέσω της νομοθετικής διαδικασίας. Μετά για το ερώτημα της κυρίας Κώστα. Αρχικά είπατε για την ε, σύγκριση ε, μεταξύ νεότητας και αθλητισμού. Έχετε δίκιο, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στον αθλητισμό καθόλου. Θέλουμε να υπάρχει όμως ισότιμη μεταχείριση. Αν τώρα ο αθλητισμός έχει λάβει συγκεκριμένο άρθρο στη Νέα Συνθήκη που μιλάει για αρμοδιότητες και καθήκοντα και ε, λαμβάνει και συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό είπαν και οι Ιταλοί συνάδελφοι, ότι συνήθω αυτό συμβαίνει δηλαδή με τα άρθρα. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για την νεότητα. Γιατί εμεί δηλαδή δεν παίρνουμε ξεχωριστό πρόγραμμα. Η ίδια νομοθετική λογική ακολουθείται. Το ιδανικό για μας λοιπόν θα ήταν να έχουμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα Youth in Action, όχι εξαιτία ε, τη διαμόρφωση του συστήματο, όπω είπε ο κ. Μπέκερ, αλλά επειδή θεωρούμε ότι αν μέχρι τώρα το τα, το πρόγραμμα Youth in Action έχει αποδείξει την αξία του και έχει αποδείξει ότι είναι αυτό που βρίσκεται στο, ίδιο, στο ύψος των περιστάσεων και αντιμετωπίζει προκλήσεις και κρίσεις όπως πέρυσι στην Νορβηγία και φέτος στη Γαλλία. Το πρόγραμμα Erasmus δεν τα επιλύει αυτά τα προβλήματα εμείς, τα επιλύουμε ή τουλάχιστον ασχολούμαστε με αυτά. Προ το παρόν, λοιπόν, θέλουμε τουλάχιστον να έχουμε μια ανεξάρτητη γραμμή προπολογισμού. σω με κάποια άλλα ζητήματα να επιληθεί και αυτό το θέμα. Ε, για τα μίντια και πάλι αυτό θα πρέπει να επιλύσουν εκείνοι που συμμετέχουν άμεσα, δηλαδή οι οργανώσεις ε, νεότητας. Εσεί εδώ μιλάτε για τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, τα κοινωνικά μέσα ε, και την ενίσχυση της διακυβέρνηση. Βεβαίως και οι νέοι θα πρέπει να συμμετέχουν, αλλά θα πρέπει και να τους εκπαιδεύσουμε για το πώς θα ε, πρέπει να συμπεριφέρονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γι' αυτό απαιτείται και ένα πρόγραμμα που θα ενισχύει και τον, τη δημιουργική πτυχή. Για τις τρέχουσες δομές ε, και την αυτονομία, βεβαίως και συμφωνώ με όλα αυτά. Και μετά άλλο, άλλο ένα ερώτημα τη ε, Ιταλίδα συναδέλφου για τι υποτροφίε, εμεί, ω Youth Forum δεν ε, ασχολούμαστε με μόνο με αυτό, αλλά ενώσεις ε, μέλη μα. Με ενημερώνουν ότι ε, δεν είναι τεχνικό τεκμηριωμένο. Οι φοιτητέ ε, είναι αντίθετοι, λένε ότι τα κράτη-μέλη προ το παρόν ε, έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα και όχι να δημιουργήσουμε ένα ανώτερο επίπεδο γιατί αυτό προκαλεί σύγχυση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν την ευθύνη για την ε, μεταφορά και κινητικότητα των υποτροφιών. Αλλιώ τα πράγματα μπερδεύονται. Και τέλο για την στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεότητα. Και αυτό ήταν το δικό μα ε, ζήτημα, γιατί δημιουργούμε προγράμματα που αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Εμεί δεν είμαστε κατά τη πολιτική για το 2020, είμαστε υπέρ, αλλά μην ξεχνούμε ότι στην νεότητα στο συγκεκριμένο αυτό τομέα έχουμε στρατηγική. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό να τα συμφιλιώσουμε αυτά τα δύο, να τα συγκεράσουμε, αλλά στον τομέα της νεότητας έχουμε αντιλήσει σημαντικά διδάγματα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να εξηγούμε καλύτερα τι ακριβώς κάνουμε. Γι' αυτό και αρχίσαμε να μιλάμε για απασχόλησιμότητα και να εστιάζουμε την προσοχή μας στι δεξιότητες που αναπτύσσουμε. Δεν είναι η κύρια μας αποστολή, αλλά είναι ένα θετικό αποτέλεσμα της δουλειά μας, το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε. Γι' αυτό και ζητούμε από τους ε, ε, πολιτικούς εκπροσώπους ε, να διασφαλίσουν ότι όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Βούτη. Äh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για τη λεγόμενη αλλαγή παραδείγματος, υποδείγματος. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δύο προσεγγίσεις. Να κρατήσουμε τη δομή κατά δράσης αλλά να κρατήσουμε και την δομή κατά τομής. Η μία δίνει οριζόντιες γραμμές, η οποία οδηγεί σε κάποιο streamlining, σε κάποια απλοποίηση για τη διαχείριση οι τομεί όμως εξασφαλίζουν μια εμβάθυνση σε, επίπεδο πολιτικών και την καλύτερη προσαρμογή των δράσεων αυτών για τους ε, δικαιούχου. Κανείς δεν έχει πρόβλημα να υπάρξει μια, ένα επιστέγασμα που να καλύπτει, μια αιγίδα που να καλύπτει όλους αυτούς τους τομείς και όλες τις ενέργειες. Τώρα, τα νέα στοιχεία που βρίσκονται στο πρόγραμμα Εράσμου, τι μπορεί να γίνει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια, ένας εξυγχρονισμός. Έχουμε ξεκινήσει πριν από 25 χρόνια. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή προς τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνια. Έχετε δύο κύκλους, το Bachelor και το μάστερ. Αυτό προς το παρόν στο πρόγραμμα Έρασμος δεν γίνεται. Ε, δεν ακολουθείται, δεν υπάρχει υποστήριξη ιδίως στον τομέα του μάστερ. Θα πρέπει τώρα τους εκπαιδευτικούς τους διδάσκοντες που είναι οι πολλαπλασιαστέ να τους ενισχύσετε πολύ περισσότερο από τότε στο παρελθόν και θα πρέπει να σκεφτείτε καλύτερα και την διεθνή ε, διάσταση. Για τη Γερμανία, για κάθε πανεπιστήμιο η διεθνής διάσταση με την τωρινή χρηματοδότηση αφορά μονάχα ένα ή δύο άτομα η δυνατότητα δυνατοτητα ανταλλαγή. Για τη διαχείριση πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει μετά από την ε, απλοποίηση να κάνει κάποια περισσότερη επεξεργασία. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και θα πρέπει να έχουμε και λιγότερες εξετάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς. Οχτώ έλεγχοι, οχτώ δοκιμασίες γίνανε στη δική μου υπηρεσία στη Γερμανία για να ελεγχθούν τα αποτέλεσματα και παρόλα αυτά ήταν πάντα καλά τα αποτέλεσματα. Μπορεί να κάνει κανεί και λιγότερε τέτοιε δοκιμασίε για τη χορήγηση δανείων. Εδώ πρέπει να είναι σαφή τα πράγματα αυτά. Θα πρέπει να είναι συμπληρωματική αυτή η δυνατότητα με άλλες μορφές χορηγήσεων ή χρηματοδότησης. Επίσης τώρα, θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση για το Masters και για το Bachelor. Στην περίπτωση του Masters μπορούμε πράγματι να δώσουμε ένα σύστημα με δάνεια το οποίο σημαίνει και ανάληψη κινδύνου. Και θα υπάρχει και η δυνατότητα να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο να μην τελειώσει κάποιο το πτυχίο του. Αυτά λοιπόν και νομίζω μπορώ να σταθώ εδώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Ευχαριστώ πολύ δεν υπήρχαν πραγματικά απευθεία ερωτήσεις για μένα, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες για να επαναλάβω ένα σχόλιο που ακούστηκε ήδη. Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της προσέγγισής μας στη νέα πρόταση και στο νέο πρόγραμμα εξηγείται με την προέλευσή μας, εξαρτάται από το πού προερχόμαστε. Η Φιλανδία είναι μια περίπτωση όπου όλα ήδη υπάγονται σε έναν ενιαίο εθνικό φορέα και όπου υλοποιούμε ήδη το πρόγραμμα διαβίου μάθησης σαν να είχε σχεδόν όπως προτείνεται εδώ. Γι' αυτό πολλά από αυτά που είπα ισχύουν και εδώ. Συμφωνώ επίσης με τον δόκτορα Βούτιχ που λέει ότι το πρόγραμμα θα είναι καλύτερο όταν το εφαρμόσουμε από ό,τι φαίνεται τώρα πάνω στο χαρτί. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Από τη δική μας οπτική, ασφαλώς, μία από τις κυριότερες ιδέες, προσδοκίες, είναι να διαμορφώσουμε σωστά τη γενικότερη εικόνα. Να συμπεριλάβουμε όλα τα προγράμματα που πρέπει και να αντλήσουμε τα διδάγματα ε, της κοινή πείρα από τα προγράμματα που έχουμε ήδη υλοποιήσει. Τουλάχιστον στη δική μου χώρα θα επωφεληθούμε τώρα από ένα πρόγραμμα που επιτρέπει πιο εγκάρσιες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, συνεργασία με τους νέους. Ε, τι εννοώ. Ε, θα έχουμε εργαλεία μέσα, αν θέλετε, τα οποία θα μας επιτρέψουν να συνδυάσουμε την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση με τα προγράμματα νεότητας, με τα προγράμματα για την ε, νεολαία. Κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να είχαμε είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν μπορούσαμε να έχουμε έτσι μια οριζόντια προσέγγιση, εγκάρσια προσέγγιση στα πράγματα. Τώρα θα την έχουμε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επειδή δεν είμαι μονάχα πρόεδρος, αλλά επειδή είμαι και εισηγήτρια για αυτό το πρόγραμμα, και έχω σκεφτεί πάρα πολύ για πολύ καιρό για τα θέματα αυτά και έχω κάποιες ισχυρές πεπιθήσεις. Νιώθω ότι με έχετε, έχετε ενισχύσει τις απόψεις μου. Βέβαια η Φιλανδία δεν είναι η Γερμανία, δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει μια εθνική υπηρεσία στην ε, Φιλανδία με μια στη Γερμανία. Στη Φιλανδία έχει νόημα να έχει μια τέτοια υπηρεσία, τέτοιο φορέα. Στη Γερμανία όχι. Γιατί θα πρέπει ο φορέας αυτός να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο στο οποίο θα ασχοληθεί. Ο έρασμος είναι στην ΤΕΑΝΤΕ ε, μέσα στη Γερμανία. Επομένως είναι ένα κομμάτι της παιδαγωγικής ανταλλαγής σπουδαζόντων. Η κάθε χώρα λοιπόν πρέπει να έχει τη δική της δομή. Δεν πρέπει όμως να ξεπερνάει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο. Θα ήθελα τώρα μετά από όλα αυτά να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν και μετά θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Έχετε το λόγο, κύριε Κοσέτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και να ευχαριστώ σε όλους τους εμπειρογνώμονες, η συμβολή των οποίων υπήρξε και έντονη και σαφής. Θα ήθελα να πω ότι είμαι όσο ευτυχής όσο και εσείς, κυρία Πακ, γιατί και εγώ νιώθω δικαιωμένος από αυτά που υπόθηκαν. Πιστεύω ότι καταλαβαίνω ότι ακούω, κατανοώ. Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε πολλά. Συμμεριζόμαστε, για να αρχίσω, ε, την αφετηρία. Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά που είχαμε μέχρι τώρα ήταν φανταστικά προγράμματα το Youth in Action, το Erasmus Mundus, το Tempus λοιπά, Όλα αυτά είναι καλά προγράμματα. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί σημαίνει ότι χτίζουμε πάνω σε γερά θεμέλια, χτίζουμε πάνω σε κάτι που έχει αποδείξει την αξία του ως μοντέλο. Δεύτερον, ε, κάτι πάνω στο οποίο συμφωνούμε όλοι πιστεύω είναι η αναγνώριση του ζωτικού ρόλου της εκπαίδευσης, ε, της κατάρτισης και της νεότητας για την ευεξία και την ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Και νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τρίτον, ε, τρίτο σημείο συμφωνίας, σύμπτωσης απόψεων. Όλοι έχουμε υψηλές φιλοδοξίες για τις προτάσεις μας. Και τέλος, θα ήθελα να πω και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πάνω σε αυτό επίσης, ότι ε, αντιμετωπίζουμε δύσκολους καιρούς. Και για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλουμε μια πρόταση, ένα τελικό προϊόν ε, ως Επιτροπή και, και το τελικό προϊόν που θα αποφασιστεί από το Κοινοβούλιο ε, και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει αντίκτυπο σε αυτούς που λαμβάνουν απόφαση για τον προϋπολογισμό. Τα κύρια στοιχεία αυτής της πρότασης θα πρέπει να είναι πιστικά όταν θα ξεκινήσουν ε, οι έντονες συζητήσεις που θα λάβουν ε, χώρα για την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Καταρχήν, πρέπει να υπάρξει εντονότερο σύνδεσμος μεταξύ των προγραμμάτων και των χαρακτών πολιτικής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα ευθυγραμμίζονται και συμβάλλουν στους στόχους του 2020. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα ευθυγραμμίζονται και υπηρετούν του στόχους ε, της πληροφορικής για το 2020 και του ET και επίση ε, του στόχους της συνεργασίας στον τομέα της νεότητας. Και αυτό είναι θεμελιώδες. Στη συνέχεια, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα, ε, θα δώσουμε την έμφαση στα αποτελέσματα, να έχουμε έναν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Το είπε και, το είπε και ο εκπρόσωπος του Youth Forum. Και τέλος, χρειαζόμαστε απλοποίηση, όχι για μας, ούτε για τα ευρωπαϊκά όργανα, ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω ότι η Ευρωπα... Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα υπόλογο σώμα και όταν υλοποιούμε προγράμματα, στη συνέχεια πρέπει να έρθουμε μπροστά στο Συμβούλιο, μπροστά στο Κοινοβούλιο και να δώσουμε εξηγήσει ε, για την υλοποίηση των δράσεων. Αλλά φυσικά δεν είναι για μας που πρέπει να γίνει απλοποίηση. Αλλά για τους Ούτε για τους εθνικούς φορείς, αλλά για τους τελικούς δικαιούχους. Για αυτούς πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Αυτή είναι η τομή σύγκλησης, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που συμπεραίνουμε εμείς ως Επιτροπή είναι το εξής ότι παρά την επιτυχία των υφιστάμενων προγραμμάτων, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια. Κάποιοι ανέφεραν μεταβολή παραδείγματος. Πραγματικά υπάρχει αλλαγή παραδείγματος και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σε όλους τους τομείς του πληθυσμού και της νέότητα συμπεριλαμβανόμενης. Πρέπει να δούμε την αλλαγή, να, να αγκαλιάσουμε την αλλαγή αυτή και να προσαρμοστούμε. Για το λόγο αυτό θέσαμε και ε, υποβάλαμε κάποιες προτάσεις. Προτάσεις για τη βελτίωση των ήδη καλών προϊόντων μας. Βελτίωση όμως. Οι προτάσεις αυτές είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Δεν είναι όμοιες. Ε, υπάρχουν διαφορές στη νομική βάση, ε, στις ε, επεξηγήσεις που, που δείχνουν ποια, ποια είναι η σκοπιμότητα των προτάσεων της Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Να αναφερθώ σε μερικές. Πιστεύουμε ότι για να ενισχύσουμε τις συνέργειες με άλλα προγράμματα, πρέπει να αποκλείσουμε από το Erasmus for All τα άτομα που ήδη βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που είναι πιο αρμόδιο. Πιστεύουμε ότι η κινητικότητα, η οποία έχει ένα πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα και στο άτομο και στο, στα ιδρύματα και στα συστήματα, έχουν αυτόν τον αντίκτυπο μόνο όταν αυτή η κινητικότητα, είτε είναι ΒΕΤ είτε είναι άλλη κινητικότητα, ε, Α, ε, πρέπει, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να επεκταθεί στα σχολεία και στους ενήλικες. Και τέλος, έχουμε προτείνει να συμπεριλάβουμε όλα τα διεθνή προγράμματα της ανώτατης εκπαίδευσης εδώ. Πιστεύουμε ότι αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση σημαντική απλοποίηση. Ωστόσο, αυτό που έχουμε προτείνει και που έχουμε πει μέσα... Αυτά είναι, αυτές τις προτάσεις έχουμε κάνει. Ωστόσο, δεν προτείναμε κάποια από τα πράγματα που ακούστηκαν εδώ σήμερα. Δεν έχουμε προτείνει να μην αναφερθούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεότητας. προτείνουμε να κάνουμε παραπομπή. Το άρθρο 4 της προτάσης δίνει πραγματικά ε, κατευ, κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα της νεότητας. Δεν έχουμε προτείνει να μην αναφερθούμε στο Youth World, στο, στο, στον όρο νεότητα. Φυσικά, στο άρθρο 2 υπάρχει ο όρος νεότητα. Δεν έχουμε προτείνει μη συμμετοχή στην παραγωγική ζωή. Υπάρχει στο άρθρο 5 ο συγκεκριμένος στόχος και δεν έχουμε προτείνει ε, να αποκλείσουμε τα προγράμματα για τον αθλητισμό. Όλα αυτά είναι πολύ σαφή. Όταν αφορά τα σχολεία, δεν νομίζω ότι έχουμε προτείνει να το λήξουμε το θέμα. Αντίθετα, είναι χρήσιμο εργαλείο. Προτείνουμε να, αυξήσουμε την ορατότητα. Και κάτι άλλο. Ο, ο, η χρήση του όρου στρατηγική ε, συνεργασία, στρατηγική σύμπραξη. Ε, και δεν είναι ο λόγος εδώ για το μέγεθος δεν είναι ανάγκη να είναι μια τεράστια συμμαχία, μια τεράστια σύμπραξη, ωστόσο είναι στρατηγική. Επιφέρει αλλαγή. Δεν πρέπει να παρανοούμε το περιεχόμενο του όρου στρατηγική, να μην το συχαίουμε τον όρο στρατηγικός με τον όρο μεγάλος. Τα σχολεία λοιπόν και οι σχολές δεν πρέπει να φοβούνται την πρόταση αυτή. Ο κύριος Βούτιχ προτιμά για παράδειγμα ε, και την παρουσία της Ασίας και η Ασία θα βρίσκεται εκεί. Θα υπάρχει αυτή η γεωγραφική προτεραιότητα. Αναφέρθηκε επίσης στα κοινά PhDs, ε, στα κοινά διδακτορικά, στις, στις κοινέ διατριβές. Ε, δεν θα, θα, υπάρχει και αυτό, κυρίως στο Μαρία Κυρί. Στο Μαρία ε, επίσης, συμφωνώ με τον κύριο Σάλσμπερκ δεν ξέρω αν το ανέφερε εγκομιαστικά ή όχι, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε ότι και η διαβίου μάθηση συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα, όπως αναφέρατε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση και πρέπει να εξακολουθήσουμε. Η πρόταση λοιπόν πραγματικά υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτό υπόθηκε από πολλούς ειδικού εδώ και από βουλευτές που συμμετείχαν στη συζήτηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ τυπικής, άτυπης και, και ανεπίσημης εκπαίδευσης. Είναι όλα πρόσωπα του ίδιου νομίσματος και πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ενιαία προσέγγιση. Εδώ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα έγινε μια συζήτηση για το πρόβλημα της ανεργίας των νέων και αναφέρθηκαν δύο εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Και φυσικά αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα Λεωνάρντο Νταβίντσι και φυσικά και στο ε- Εράσμους. Ας το δούμε για να καταπολεμήσουμε την εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης ε, σημαίνει ότι τη, ε, προωθούμε και τη συμμετοχή στη δημοκρατία και στην ε, δημιουργία νέων που λαμβάνουν ενεργό μέρος στην κοινωνία μας. Πραγματικά αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι η σωστή. Και πιστεύω ότι ε, μόνο με ολιστική προσέγγιση θα επιτύχουμε συνέργειες. Στη συνέχεια, κάτι που δεν έχουμε προτείνει είναι να ανταγωνίζονται οι διαφορετικοί τομείς μεταξύ τους. Δεν το προτείνουμε αυτό. Ασφαλώς Ασφαλώς, οι κοινοπραξίες των Ιδρυμάτων Ανωτά Εκπαίδευσης για να αντιμετωπίσουν το δύσκολο αυτό καθήκον της δημιουργίας ενός κοινού μάστερς. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να έρχεται σε ανταγωνισμό με ένα άτυπο δίκτυο ε, νέων εργαζόμενων. Ούτε με τα δίκτυα των σχολείων, ούτε με τα δίκτυα των σχολών, ούτε με άλλες μορφές συνεργασίας. συνεργασίας. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και γι' αυτό ε, στην, στο μήνυμά της ε, που συνοδεύει την ε, νομική βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά μιλά για τις ελάχιστες συνεισφορές ανατομέα. Αυτό είναι βασικό, ζωτικό. Νομίζω ο κύριος ανέφερε ότι έχουμε την πραγματικότητα και η πραγματικότητα δεν μπορεί να αναχθεί σε μια τρισέλιδη ανακοίνωση. Αυτό που δεν ε, Μόνο η, προσέγγιση, μόνο η εξορθολογήκευση, μόνο ο τρόπος προσέγγισης του πράγματος. Αλλά βέβαια η πραγματικότητα υπάρχει εκεί και φυσικά θέλουμε να έχουμε αντίκτυπο στην πραγματικότητα ε, για να επιτύχουμε και τους στόχους για το 2020 για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας στην Εκπαίδευση και στην Νεότητα. Όλα αυτά πρέπει να είναι πολύ σαφή. Και κάποια τελευταία πράγματα πάνω στον τίτλο. Το, ο τίτλος Erasmus for All, το πρόγραμμα Erasmus για όλους, είναι ο σωστός τίτλος. Ο όρος Εράσμους είναι πασίγνωστος. Όλοι ξέρουν ότι συνδέεται με, με τη λέξη αυτή η νεολαία, η κινητικότητα. Όλοι γνωρίζουν τι είναι το Εράσμους. Και η, κυρία Πρόεδρος το είπε, ότι πολλοί όταν θέλουν να αναφερθούν στα προγράμματα ε, όταν θέλουν να αναφερθούν στην κινητικότητα και να κάνουν κάτι για την κινητικότητα, θέλουν να συνδεθούν με τα προγράμματα έρασμος. Και φυσικά αυτό είναι σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο στην ανώτατη εκπαίδευση εστιάζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο η απασχολησιμότητα μας απασχολεί. Ότι όλα τα άλλα τα έχουμε λησμονήσει. Ότι οι άλλοι στόχοι έχουν λησμονηθεί. Καλύτερο είναι να πούμε όμως Erasmus for all και όχι all for Erasmus. Και όχι ο, ο για όλους και όχι όλοι για τον Ερασμό». Είπατε ότι όταν δούμε τον προπολογισμό τότε θα, αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τον προπολογισμό. Κυρία Πάκο όμω, ε, φυσικά καταλαβαίνετε ότι πρέπει η πρόταση που θα υποβάλουμε να είναι η υγιής και αξιόπιστη όχι μόνο για μας εδώ. Εδώ ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των κέντρων νεότητας, αλλά σε, σε άλλες αίθουσες, σε άλλα φόρα ε, που, που κάθονται άλλοι αρμόδιοι επί άλλων ζητημάτων, εκείνοι δεν γνωρίζουν για αυτά. Δεν γνωρίζουν τι είναι χρήσιμο για μας. Πρέπει να, τους, πρέπει να υποβάλουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που να καλύπτει όλα αυτά που είπαμε. Πρέπει να παρουσιάσουμε λοιπόν κάτι όμως πιστικό για τους Υπουργούς Οικονομικών, οι οποίοι στο τέλος θα υπογράψουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κορέλ. Δεν πρόκειται τώρα να πω όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε στην Επιτροπή μας και ακούσαμε στην ακρόαση. Κύριε Κορέλ όμως, αλλά νιώθω κάποια ανησυχία όταν προσπαθώ να, όταν πρέπει να προσπαθήσω να καταλάβω τι ακριβώς εννοείτε. Πού είναι αυτά λοιπόν που λέτε ότι υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική εικόνα. Δεν έχουμε λοιπόν μια τέτοια πραγματική σαφή εικόνα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμάτε το κοινοβούλιο. Εγώ και οι συνάδελφοί μου έχουν εκλεγεί για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς στόχους. Δεν έχω εδώ πέρα εκλεγεί για να δίνω εξηγήσει σε μη εκλεγμένους διοικητικού υπαλλήλου. Έχετε κάνει μια πρόταση, συζητήσαμε για το θέμα αυτό, φέραμε εδώ εμπειρογνώμονε και νομίζω ότι όλοι έχουμε την άποψη ότι χρειαζόμαστε μια, ένα συνδυασμό της καλής σας πρότασης τουλάχιστον σε μένα φαίνεται καλή πρόταση των ε, δράσεών σας συνδυασμό με μια κατατομής οργάνωση, ώστε να ξέρει ο καθένας ποια είναι τα δικά του κουκιά και ποια είναι των άλλων. Εμείς δεν ξέρουμε, όπως είναι τώρα τα πράγματα, τι θα πρέπει να δώσουμε για το Εράσμους, το οποίο ήταν ένα κοινοτικό πλαίσιο για τους φοιτητές και τι θα δώσουμε για τους μαθητές των σχολείων. Το κομμένιος είναι μια κοινότητα ανθρώπων, το Γκρούτφιχ είναι μια κοινότητα ανθρώπων. Θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι υπεύθυνοι της Κομισιόν. Δεν μιλάω για σας προσωπικά. Είναι ωραίος λοιπόν ο έρασμος και ε, όλοι το καταλαβαίνουν. Μα όταν καταλάβει κανεί τι σημαίνει ο έρασμο στο καινούριο τρένο, θα πει τρελή είναι αυτή τώρα. Θέλω να τα βάλω όλα αυτά εκεί πέρα. Αυτό για τα ονόματα, δηλαδή το όνομα Εράσμους για όλους, υπόσχεται κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο θέλετε εσείς να πετύχετε, το θέλουμε και εμείς κύριε Κόρελ. Ήμουνα εισηγήτρια στα θέματα αυτά ήδη από το 1992. Είπαμε ότι η διαβίου εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η βασική έννοια και κάτω από αυτή την στέγη έχουμε διάφορους τομείς οι οποίοι θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Δεν τα καταφέρατε τα τελευταία πέντε χρόνια να τους συνδέσετε. Δεν φταίμε εμείς. Και τώρα θέλετε να τα κάνετε όλα εράσμους και να αφήσετε τα άλλα προγράμματα. Είσαστε ο συνομιλητής μας κύριε Κορέλ, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να απευθυνθώ σε εσά. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μια τακτική διαδικασία, μια οργανωμένη διαδικασία και χρειαζόμαστε κατευθύνσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε κάτι το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε αυτά τα οποία λέτε. Αν εσείς καλύπτετε το 56% με αυτές τις δράσεις από ό,τι υπολόγισα, τι κάνετε με τα υπόλοιπα 44%. Δεν μπορώ να σας δώσω περιθώριο ελιγμών 44%. Το κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών το 44%. Άντε 10% μπορώ να σας δώσω αν θέλετε να έχετε περιθώριο. Τα άλλα 90% όμως θα πρέπει να κατανεμηθούν στους διάφορους τομείς. Και σίγουρα πρέπει να κάνουμε πράγματα για την κινητικότητα, την συνεργασία κτλ. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ποια είναι τα αριθμητικά ποσά τα οποία συνδέονται με κάθε τομέα και κάθε δράση. Αυτή τη στιγμή είναι λιγάκι ανακατεμένα. Εμείς ακούσαμε προσεκτικά λοιπόν τις απόψεις σας και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα το κοινωνικό ταμείο στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει Λεωνάρντο Νταβίτσι που έχει κάποιους τομείς εκεί. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ατόμων που είναι μακροχρόνια άνεργοι. Μπορεί να βοηθήσει αυτούς που θέλουν να κάνουν μια μαθητεία σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, μαζί σας θέλουμε να έχουμε μια στρατηγική συνεργασία στον τομέα αυτό, αλλά για το Κομένιους εγώ συμφωνώ <clears throat> απόλυτα με τον εκπρόσωπο, με τον ομιλητή προηγουμένως. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε στα σχολεία δεν ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική για φέτος. Όταν είναι έτοιμη να ετοιμάσουν κάτι οι διδάσκοντες θα πρέπει να ξέρουν πάνω σε τι βασίζονται. Δεν είσαστε εσείς που έχετε την ευθύνη για τα σχολεία, ούτως ή άλλως. Είναι οι διδάσκοντες οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν για το πρόγραμμα. Λοιπόν, η στρατηγική είναι μια καλή ιδέα, αλλά τα σχολεία θα πρέπει να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες και εγώ χαίρομαι όταν οι δάσκαλοι είναι σε θέση να τα κάνουν αυτά. Ο στόχος είναι σαφής. Ο στόχος είναι να γίνουν Ευρωπαίοι οι μαθητές. Και τώρα ο κύριος Στάκουλα έφυγε που θα, τα, θα σας τα έλεγε και αυτός. Το κομμένιος δεν είναι για τους διδάσκοντες, είναι για τους μαθητές. Θέλουμε όμως και οι δάσκαλοι να έχουν τη δυνατότητα μετεκπαίδευση και αυτό να είναι κομμάτι του προγράμματος αυτό. Το έχω πει πριν από τη νέα προγραμματική περίοδο στην Κομισιόν και φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει η Κομισιόν αυτό. Σας ζητώ λοιπόν να το σκεφτείτε και τέλος υπενθυμίζω στην Κομισιόν ότι η ιδέα του κομμένιου Σρέγγιο ήταν δικιά μου ιδέα. Το εδέχθη η Κομισιόν και είναι κάτι το οποίο λειτουργήσε πολύ καλά σε πολλούς τομείς. Γιατί λοιπόν αυτή η ιδέα να μπορέσει να λειτουργήσει σε ένα τομέα και όχι, όχι. Πάρτε την ιδέα του κομμένου Ρέγκερ και επεκτείνετε και στον άλλο χώρο. Κάντε μία προσέγγιση και κατά και εγώ είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε από κοινού να επιτύχουμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις ιδέες. Και εντάξει, κάπου πρέπει να βγάλω και την αδρεναλίνη μου και γι' αυτό σας μιλάω μερικές φορές επικριτικά και έντονα. Νομίζω ότι με αυτή τη συνεργασία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι και θα ήθελα να πω και στον εκπρόσωπο των νέων για τα προγράμματα των νέων. Εγώ έχω συζητήσει με πάρα πολλούς. Αν θέλω να έχω ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα για τους νέους, θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι έχει μια θέση στο συνολικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τους νέους, αλλά αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς, θα πρέπει να έχει και το δικό του προϋπολογισμό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία με καίγανε και τα όλα αυτά τα οποία με είχαν οδηγήσει να αγωνιστώ όταν ήμουν πιο νέα, σας τα έχω βγάλει σας ευχαριστώ λοιπόν όλους τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ και την Κομισιόν και σας εύχομαι να έχουμε μια καλή συμφωνία η οποία μπορεί να προκύψει από τις προτάσεις της Κομισιόν. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε μια καλύτερη λύση για το καλό όλων. Ευχαριστώ. Τέλος της συνεδρίας.